Dear friends, ladies and gentlemen, let's start. We have uh, the agenda here. Καλησπέρα, έχουμε την ημερήσια διάταξη. Λοιπόν, το θέμα για τη Λετωνία θα πρέπει να συζητηθεί και κλεισμένο των θυρών. Θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Ε, για να γίνει αυτό γύρω στις 5.30. Θα ήταν δυνατόν σε μία ώρα πρέπει να φύγω με κάποιους σοσιαλιστές και φιλελευθέρους. Ε, λόγω των διαπραγματεύσεων στο Κίσιναου, είπαμε, Λοιπόν, μπορούμε να συζητήσουμε κάποια θέματα σήμερα το απόγευμα. Τις ε, εκθέσεις για τα Βαλκάνια. Ίσως αύριο το πρωί ε, μπορεί κάποιος από τους συναδέλφους να συζητήσει αυτή την έκθεση αντί τη δική μου. Δεν έχουν φτάσει όλοι οι συνάδελφοι. Μπορούμε λοιπόν κάτι να κανονίσουμε. Είναι σημαντικό όμως το ταξίδι βλέπετε αύριο να πάμε στην χώρα εκείνη. Έγκριση των πρακτικών. Έχετε κάτι. Δεν υπάρχει παρατήρηση. Ανακοινώσεις του Προέδρου δεν έχω τίποτα. Να δούμε κατά πόσο το έγγραφο για το Συμβούλιο Γιατί η Ρωσία που είναι άτυπο και το έχουν όλοι. Τι είναι αυτό, τι γίνεται. Μπορούμε και εμείς να το έχουμε. Μπορεί να διανεμηθεί στα μέλη ίσως να βοηθά τις συζητήσεις για τη Λετωνική Προεδρία που θα γίνει στις 5.30. Αν μπορούν να το τυπώνουν και τα μέσα ενημέρωσης μπορούμε να δείξουμε το έγγραφο αυτό και στα μέλη της Επιτροπής μας. Θα είναι και ένα από τα σημαντικά θέματα της συζητήσεως των Υπουργών Εξωτερικών. Εκθέσεις προόδου Α, έφτασε ο συνάδελφο αρμόδιο. Τσαλ Τάνοκ. Α, αύριο. Τσαλ, μπορείς αύριο. Είσαι φίλος μου. Ο κ. Μακάλιστερ, Σερβία. Καλησπέρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι τιμή για μένα να παρουσιάσω το σχέδιο ψηφίσματος για την έκθεση πρόοδου του 2014 για τη Σερβία. Δεν είναι μόνο το πρώτο σχέδιο κειμένου του συγκεκριμένου ψηφίσματος, είναι και πρώτο μου έγγραφο σαν μόνιμος συντονιστής, σαν μόνιμος εισηγητής για τη Σερβία. Λοιπόν, επισκέφθηκα τη Σερβία τον Νοέμβρη, πες για μια εβδομάδα συνάντησα τον Πρωθυπουργό Βούτσιτ, τον κύριο Τάτσον Υπουργό Εξωτερικών, τον Πατριάρχη Ειρηνέο, μέλη της και κυβερνητικέ οργανώσει, εκπροσώπου του οικονομικού τομέα, τη κοινωνία των πολιτών. Πολλά πράγματα άκουσα, πολλά παρατήρησα στο Βελιγράδι και στο Νόβισαντ που ήταν σημαντικά για την έκθεσή μου. Λοιπόν, το κείμενο έχει 24 παραγράφου και 6 σελίδε Προσπάθησα να είμαι όσο πιο ακριβής και σύντομος μπορούσα βλέποντας τι έγινε το 2014, τη σημαντικό για τη Σερβία, ε, ξεκίνησαν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις επισήμως στις 21 Ιανουαρίου στην πρώτη διακυβερνητική διάσκεψη Ευρωπαϊκής Ενώσεως Σερβίας. Η τεχνική ανάλυση έχει δρομολογηθεί και ήδη έχει ολοκληρωθεί ε, για 26 κεφάλαια. Το υψηλό επίπεδο προετοιμασίας και η εξέταση εφαρμογής ε, του κοινοτικού κεκτημένου ε, είναι κάτι επί το οποίο κινήθηκε σωστά η Σερβική κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργό Βούσιτ και η κυβέρνησή του ε, θέλουν να πετύχουν στην ενταξιακή αυτή πορεία και θέλουν να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά προβλήματα, να κάνουν τι αναγκαίε μεταρρυθμίσει. Πρόσφατα η Σερβία θέτησε σημαντικέ ε, σημαντικούς νόμους για τα εργασιακά, για την ενημέρωση, ιδιωτικοποίηση, για την χρεοκοπία, για τους πληροφοριοδότες κλπ. Και όλα αυτά είναι σημαντικά. Χρειάζεται διεξοδική όμω εφαρμογή τη νομοθεσία και των διαφόρων πολιτικών. Και αυτό θα δείξει κατά πόσο η όλη ε, διαδικασία ήταν επιτυχής. Να τονίσω τέσσερα πράγματα. Πρώτον, το κράτο δικαίου. Η σερβική κυβέρνηση έχει θέλει να προσπαθήσει να καταπολεμήσει τη διαφθορά, όμως χρειάζονται σημαντικές προσπάθειες για να εφαρμοστεί το κατάλληλο νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Και κάτι άλλο, να τονίσω τη σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων της αντιπολιτεύσεως. Τώρα πάρα πολλοί νόμοι υιοθετούνται ε, στα πλαίσια της κατεπίγουσας ανάγκης που δεν επιτρέπει ε, στους εμπλεκόμενους φορείς να εκφράσουν τις απόψεις τους. Έτσι δε περαιτέρω, μίλησα με παρατηρητές στο Βελιγράδι και ανησυχούν για την επιδείνωση της καταστάσεως όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης στη Σερβία και υπογραμμίζω ότι η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης είναι βασικό στοιχείο της δημοκρατίας. Δεύτερον, η οικονομία θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τη σερβική κυβέρνηση και τις σερβικές αρχές να προβούν σε περαιτέρω διαθροτικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις για να βελτιωθεί το κλίμα για τις επενδύσεις, να καταπολεμηθεί το υψηλό επίπεδο της ανεργίας και να συνεχινιστεί η οικονομική εξυγίανση. Το επιχειρηματικό περιβάλλον χρειάζεται βελτίωση μέσω εφαρμογής των στοιχειωτικών αλλαγών και μέσω ενίσχυσης του νομικού συστήματος. Όμως θα πρέπει να λάβουμε επίσης υπόψη ότι οι πλημμύρες του Μαΐου του 2014 στη Σερβία είχαν αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία και βέβαια και για τους λαούς που ζούσαν στις περιοχές της πληγήσεως. Τρίτον, εξωτερική πολιτική. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι σαφείς οι κανόνες. Οι υποψήφιες χώρες θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με το κεκτημένο το ευρωπαϊκό και αυτό ισχύει και για την εξωτερική πολιτική. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Σερβία ιστορικά έχει στενές σχέσεις με τη Ρωσία. Παρόλα αυτά, λυπούμε διότι η Σερβία δεν ευθυγραμμίστηκε όταν εκλήθη να το κάνει αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τα περιοριστικά μέτρα κατά της Ρωσίας. Από την άλλη πλευρά, καλωσορίζω θερμά το σχέδιο δράση για την ειδική σχέση μεταξύ ΝΑΤΟ και της Δημοκρατίας της Σερβίας που υπεγράφει εδώ και τέσσερις ημέρες Επίσης καλωσορίζω την Προεδρία της Σερβίας του ΟΑΣΥ το 2015. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την προνομία χαθές της Σερβίας, κυρίως όσον αφορά ε, τη Ρωσία για να βρει ε, λύσεις όσον αφορά την κρίση στην Ουκρανία. Και τέλος, τέταρτο σημείο, η εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινα. Η Σερβία θέλει να εξομαλύνει τις σχέσεις με το Κωσυφοπέδιο και αυτό είναι πολύ ευπρόσδεκτο. Λόγω των προήμων εκλογών στο σερβικό κοσυφοπαίδιο, η πορεία των διαπραγματεύσεων, ο ρυθμός διαπραγματεύσεων επιβραδύνθηκε το 2014. Γι' αυτό καλωσορίζω ότι μετά από ένα εξάμεινο πολιτικού πολιτικής αποτελμάτωσης και διαμάχης των κομμάτων, το Κοινοβούλιο του Κωσυφοπεδίου διόρισε τον κύριο Μουστάφα σαν νέο Πρωθυπουργό. Και το διάλογο υψηλού επίπεδου Σερβίας Κωσυφοπεδίου θα συνεχιστεί στις, εδώ στις Βρυξέλλες στις 9 Φεβρουαρίου. Είναι σημαντικότατο το ότι η Σερβία και το Κωσυφοπέδιο προχωρούν εφαρμόζοντας τις επιτευχθήσεις συμφωνίες. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, εν γέννη, έχει μπει στις ράγες του το τρένο από τις, ε, ε, το σερβικό προς, την, ε, προς Βρυξέλλες, το τρένο του Βελιγραδίου, να παραμείνει στην τροχιά και θα πρέπει να ανοίξουν τα πρώτα κεφάλια τα διαπραγματευτικά το 2015 Ελπίζω ε, το πρώτο εξάμεινο του 2015 να γίνει αυτό. Εν τέλει θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γραμματεία του ΕΛ και την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για την υποστήριξή της. Ελπίζω σε καρποφόρα συνεργασία μαζί σας, κυρίως με τους κοιόδους εισηγητές, ούτω ώστε τελικά να πετύχουμε καλά αποτελέσματα. Θέλω να ακούσω και τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις σας και σας ε, ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Είναι στον επόμενο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Δεν διαφωνώ σε τίποτα από όλα όσα μας εξέθεσε. Κύριος Μεκάλιστερ. It is, it is absolutely clear. Είναι ηλίου φαϊνότερον ότι χωρίς καμία αμφιβολία προχωρεί και προεδεύει η Σερβία προς την ένταξή της. Αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε και όντως το αναγνωρίστηκε σε αυτή την έκθεση και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, το πιο βασικό για τη Σερβία είναι να συνεχίσει αυτή την ε, πορεία πρόοδου. Πρόοδο στην οικονομία, πρόοδο στις γενικές μεταρρυθμίσεις. Επίσης θα πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις ε, τα κεφάλαια 23 και 24 όσον αφορά την δικαιοσύνη και αυτά θα μετρήσουν στις διαπραγματεύσεις. Επίσης θα πρέπει να χαιρετήσουμε ε, και να καλέσουμε τους εισηγητές να διαφωτίσουν τα σημεία που έχουν τη σχέση με τη Ρωσία, γιατί θα έχει η Σερβία τη μοναδική ευκαιρία να αποδείξει ότι θα μπορούσε να επιδείξει την προοδό και να την αποδείξει ε, με, όταν τρόπο θα ασκήσει την προεδρία του ΙΣΥ. Επίσης θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει η υλοποίηση όλων αυτών τα οποία έχουν υπογραφεί. Επίσης θεωρώ ότι έχουμε και το κεφάλαιο για τη σχέση με το κοσμοπέδιο και αυτό το κεφάλαιο θα πρέπει στις θέσεις διαπραγματεύσεις να ανοίξει εγκαίρως και θα είναι σημαντικό να έχει η Σερβία καλές σχέσεις με τις χώρες της ε, περιοχής. Είναι ήταν σημαντική η επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Αλβανίας ε, παρά τα όσα συνέβησαν σε σχέση με την επίσκεψη εκείνη και όπως είπα η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης είναι πάρα πολύ βασικό σημείο της πορείας προόδου και επίσης συμφωνώ με τον κύριο εισηγητή για τα όσα είπε όσον αφορά την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, το όλο κλίμα σε αυτόν τον τομέα να ε, ε, βελτιωθεί η διαφάνεια για την ιδιοκτησία, να αντιμετωπιστούν οι απειλέ κατά δημοσιογράφων. Επίση, κύριε Πρόεδρε, κάτι άλλο όσον αφορά την ε, δέσμευση των ε, χωρών των Δυτικών Βαλκανίων όσον αφορά κάποιου είδου μακρόπνε στρατηγικέ. Αυτό σα το αναφέρω σε σχέση με τα σχέδια επενδύσεων, ιδίω όσον αφορά ε, τα ενεργειακά. Ήμουνα στην συνάντηση κορυφή του, του Βελιγραδίου και είπαμε ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικά τα όσα συμφωνήθηκαν για την ενέργεια και συμφωνήθηκε ότι θα γίνουν και άλλα οπότε μια που θα έχουμε κάποιου μακρόπνε μακρόπνες επενδύσεις θα είναι σημαντικό να δούμε τι θα γίνει με αυτού του είδου τα σχέδια σε σχέση με τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είχαμε επίσης και το επεισόδιο με την Φαλονγκόνγκ, οπότε θα πρέπει να ζητηθούν κάποιε εξηγήσει, αλλά έχουμε και ε, άλλα σημεία στην έκθεση του Ντέιβιτ. Πάντως θα πρέπει να τον επενέσουμε για το πώς ασχολήθηκε με αυτή την ε, έκθεση και να του πούμε μπράβο για το αξιόλογο έργο που μέχρι τώρα έχει επιτελέσει. Ο επόμενος. Ευχαριστώ πάρα θα μιλήσω σλοβενικά και αυτό ελπίζω να είναι πιο κοντά και στους Σέρβους ε, φίλους μας. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον David Μακάλιστερ, τον εισηγητή, για την ε, εξαιρετική αυτή, σύντομη αλλά περιεκτική έκθεση. Κάποια σημεία μπορούν να βελτιωθούν περαιτέρω και είμαι πεπισμένη ότι από κοινού θα καταφέρουμε να βελτιώσουμε την ε, έκθεση. Το τελευταίο μισό χρόνο έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικά περιστατικά οι κοινοβουλευτικές εκλογές, οι υψηλόβαθμοι επισκέπτε το Βελιγράδι, η διπλωματική δραστηριότητα της Σερβίας ενισχύθηκε και στην ε, περιοχή διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο η Σερβία. Το τελευταίο έτος όμως ήταν και δύσκολο λόγω των πλημμύρων που έπληξαν τους πολίτες, τις υποδομές αλλά και την ίδια την οικονομία. Ο εισηγητής προειδοποιεί Λόγω της ε, συνεχώς ε, επιδεινούμενης κατάστασης ε, σε διαφορετικά τα μέσα ενημέρωσης, συμφωνώ με την ανησυχία του και στις διαπραγματεύσεις της πρωταξιακές δεν άνοιξαν νέα κεφάλαια. Μας λυπεί αυτό. Στην αρχή του έτους η Σερβία ανέλαβε και την Προεδρία του ΆΣΕ. Αυτό είναι κάτι που το καλωσορίζουμε. Ελπίζουμε λοιπόν το διπλωματικό δίκτυο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση των συγκρούσεων στο εσωτερικό της περιοχής του ΑΣΕ και σε ό,τι αφορά και την Ουκρανία ασφαλώς. Αυτό που με ανησυχεί ιδιαίτερω είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά τα μέσα ενημέρωσης όπως ανέφερα. Το παρακολουθώ αυτό πάρα πολύ στενά και διαπιστώνω ότι είναι όλο και μεγαλύτερη η επιδείνωση και σε ό,τι αφορά μια σύγκριση με τον καιρό του Μιλόσεβιτς. Ε, διαρκώς ε, χειροτερεύουν οι συνθήκες εργασίας των δημοσιογράφων και οι μορφές και οι δομές ιδιοκτησίας σε ό,τι αφορά τα μέσα ενημέρωσης είναι προβληματική και όπως έχει κατηγορήσει κάποια μέσα ενημέρωσης για διάδοση ψευδών ειδήσεων. Αυτά είναι όλα ανησυχητικά. Και θα ήθελα να πω ότι αυτό αφορά και τον πλουραλισμό. Αποτελεί, ξέρετε, ο πλουραλισμός αυτός ε, στην έκφραση ένδειξη μιας ε, υγιούς κοινωνίας. Δεν είναι ικανοποιητική κατάσταση στην ε, Σερβία. Μία παρατήρηση να κάνω ακόμη. για την κοινότητα, την, την ομάδα των ΛΟΑΔ. Χαίρομαι που τον περασμένο Σεπτέμβριο έλαβε χώρα το Gay Pride στην ε, Σερβία, στο Βελιγράδι. Είναι σημαντικό να τονιστούν τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στο άρθρο 14 του Σερβικού Συντάγματος. Αλλά η κοινότητα των ΛΟΑΤ θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω. Τέλος, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με το Κωσυφοπαίδιο στις 9 Φεβρουαρίου, θα γίνει προεδρική συνάντηση. διαμεσολαβητές ήταν και τα θεσμικά όργανα των Βρυξελών στον τομέα αυτό. Νομίζω ότι χρειάζεται μια ανάλυση των σχέσεων. Και κλείνοντας θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι είναι πια καιρός η Σερβία να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις πρωταξιακές διαπραγματεύσεις. Το νέο έτος λοιπόν δεν θα πρέπει να είναι μόνο δυναμικό όπως και το περασμένο έτος, αλλά και ένα έτος με πολλά νέα κίνητρα και στις πρωταξιακές διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Uh, thank you, Mr. President. On behalf ECR, e I too congratulate από το ECR να συγχαρώ τον κύριο Μακάλιστερ σε αυτή του την uh, παρθενική εισήγηση αφορά την Σερβία, πολύ καλή του η προσέγγιση και επιμελής. Η πολιτική μας ομάδα χαιρετίζει την πρόοδο της Σερβίας σε διάφορους τομείς όπως πολέμηση της διαφθοράς, μεταρρυθμίσεις, βελτίωση σχέσεων με κοσυχοπαίδιο και επίσης όπως λέει και η πρόσωπος θα συνεχιστεί ο διάλογος Πριστίνας Βελιγραδίου. Πάντως προβληματίζουμε ακόμη για το νέο άρθρο 224 ήδη οι εμπλεκόμενοι έχουν ε, παραπονεθεί σε σχέση με κάποιες απαρτριώσεις που αφορούσαν ε, το παλαιό ε, δίκτυο και συνεχίζονται. Ο κύριος Κούκαν ε, είπε ότι θα συνεχιστεί η μεταρρύψη της ε, δικαιοσύνης, ε, κατάρτιση δικαστών, ανεξαρτησία, αμεροληψία. Επίσης είναι πάρα πολύ θετικό το ότι τώρα οι σχέσεις είναι καλύτερες με το κοσυφοπαίδιο. Επίσης, όπως ότι έχω αναλάβει μόνιμο σύγκριση για το Μαυροβούνιο και εκεί έχουμε πρόοδο, έχουμε και από τις δύο πλευρές ανταλλαγή επισκέψεων και Είπαμε ότι οι φυγόδικοι ε, τώρα ε, εκδίδονται από τη μία χώρα στην άλλη για να επιληθεί η δικαιοσύνη. Επίσης, και εγώ όπως ο καλύτερα, έχω επικρίνει την προσέγγιση της κυβέρνησης Νίκολης Βούησιτς όσον αφορά τις στενές σχέσεις με την ε, Ρωσία και τα όσα έγιναν στην επίσκεψη Πούτιν στο Βελιγράδι, τις κοινέ ταξιδικές ασκήσεις τώρα που η Ρωσία έχει επιτεθεί στην Ουκρανία και έχει καταλάβει την Κρυμαία. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με τις θετικές εκτιμήσεις σε ό,τι αφορά την πρεμιέρα του κ. Μακάλιστερ ως εισηγητή. Έλαβα και τις πληροφορίες σε ό,τι αφορά τη Σερβία. Και είναι πολύ καλό το γεγονός ότι επιδεικνύει τόσο ενδιαφέρον ως εταίρος. Να υπογραμμίσω ότι σύμφωνο με τα όσα είπε ο προλαλήσαντας, ότι ο τομέας των μέσων ενημέρωσης είναι ένα πάρα πολύ ευάλωτο και ευαίσθητο ζήτημα στη Σερβία, το οποίο χρήζει βελτίωσης. Θα πρέπει να συγχαρούμε τη, τη Σερβία για μια πρώτη βελτίωση σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς, ιδιαίτερα τη διαφθορά υψηλού επίπεδου στα ανάτατα κλιμάκια. Εκφράζουμε ικανοποίηση για το γεγονός ότι η κυβέρνηση δείχνει δέσμευση στην ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας. Είναι σημαντική αυτή η αλλαγή και εξίσου σημαντικό είναι ότι η κυβέρνηση αυτή έχει μία αντιπολίτευση επίσης δεσμευμένη για το σερβικό μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο ήταν πολύ διαφορετικό στο παρελθόν. Νομίζω ότι η Σερβία θα πρέπει να αναγνωριστεί σε ό,τι αφορά την επικοδομητική της πολιτική προς τους γείτονες και για το θάρρος που έχει επιδείξει να διορθώσει κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζει με ομόρες χώρες. Θα ήθελα να καλέσω τον εισηγητή να δώσει ιδιαίτερη σημασία στη Βοηβοντίνα. ως το πλέον προηγούμενο και προευρωπαϊκό τμήμα της Σερβίας. Η αυτονομία της ε, Βοηβοδίνα είναι κάτι το οποίο εξετάζεται. Και τέλος, να συμφωνήσω κι εγώ με την ανησυχία σε ό,τι αφορά τον συντονισμό της, Ευρωπα... της πολιτικής ε, εξωτερικών υποθέσεων της Σερβίας με την ευρωπαϊκή αντίστοιχη πολιτική. Τέλος. Ε, Σε ό,τι αφορά το ΣΕΣΕΛ, καταλαβαίνω ότι ο νεοεκλεγής ε, πρόεδρος ζήτησε από το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να παρέμβει, προκειμένου το ΣΕΣΕΛ να επιστρέψει στη Χάγη. Αυτό δεν έχει να κάνει τίποτα με την σερβική κυβέρνηση και δεν θα πρέπει η σερβική κυβέρνηση να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις δηλώσεις του ΣΕΣΕΛ, αλλά νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει και με την δική μας αντιμετώπιση. Θα πρέπει να βρούμε μια λύση για το θέμα αυτό και να εκφράσουμε την απόψή μας στη συνέχεια ενδεχομένω για την απόφαση της, Δικαστήριας της Χάγης. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν ξεκινήσω να σχολιάζω την έκθεση για τη Σερβία, να πω ότι αν είχαμε το αρχικό μας σχέδιο να ξεκινήσουμε στις 3, αν ξεκινήσουμε στις 3 θα μπορούσαμε να είχαμε συμπεριλάβει και την έκθεση ε, του κυρίου Μπροκ. Αντί για να συζητήσουμε σήμερα και την ομάδα μου είναι πραγματικά δύσκολο να αναδιοργανώνουμε σήμερα τι εκθέσει σήμερα και αύριο, διότι έχουμε διαφορετικού σκιώδει για διαφορετικέ εκθέσει. Εγώ θα προτιμούσα το πρόγραμμα να είχε παραμείνει όπω ήταν αρχικά. Αυτό ήθελα να πω. Αλλά αποφασίστηκε να γίνει διαφορετικά. Για μικρότερε ομάδε όμω αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνονται την τελευταία στιγμή αλλαγές στην ημερήσια διάταξη. Ε, είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε όλες εκθέσεις επιτάπητος για τις επόμενες εβδομάδες. Διότι είναι πολύ σημαντικό το Κοινοβούλιο να στείλει ένα σαφές μήνυμα μέσω των εκθέσεων. Και στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Γιούνκερ, που πριν εκλεγεί είχε δηλώσει ότι δεν θα γίνει διεύρυνση εντός επόμενης πενταετίας ότι ξέρουμε ότι είναι μια πολιτική πραγματικότητα αυτή. Αυτό κόστισε όμως προβλήματα, μείωσε τα κίνητρα διαφόρων χωρών. Και χαίρομαι που είμαστε εδώ και λέμε το Κοινοβούλιο είναι υπέρ της συνεχιζόμενης στρατηγικής της διεύρυνσης με όλες τις χώρες της περιοχής. Για την έκθεση του κ. Μακάλιστερ. Τον ευχαριστώ και εγώ. Είναι νέος συνάδελφος που ασχολείται με τα Δυτικά Βαλκάνια, έξοχη έκθεση του. Έκανες πολύ καλή δουλειά πραγματικά και σε βασικών θεμάτων και είναι χαρά μου η συνεργασία μαζί σου. Συμφωνώ με τις θυγήσεως πτυχές. Παρ' όλα αυτά. Δεν ξέρω αν θα είναι καιρός εδώ σκιώδης μας για τη Σερβία. Είναι σε άλλη επιτροπή τώρα. Και θα ερχόταν αργότερα. Θα ήταν σημαντικό λοιπόν να συμπεριληφθούν ενεργειακές πτυχές και το περιβάλλον. Διότι οι ευρωπαϊκοί στόχοι για τις εκπομπές συνεπάγονται διαφορετική στρατηγική για τη Σερβία. Να παράγει ηλεκτρισμό, ηλεκτρική ενέργεια από άλλε πηγές και όχι από άνθρακα. Πρέπει να υποβάλουμε σχετικές τροπολογίες. Πρέπει να προσθεθούν κάποια στοιχεία. Οι σχέσεις με τη Ρωσία αναφέρονται και καλώς στην έκθεση και κυρίως οι σχέση μεταξύ Σερβίας και Κωσυφοπεδίου. Σαν εισηγήτρια για το Κωσυφοπέδιο, σε ευχαριστώ για τα σημαντικά στοιχεία παραθέτης. Καλό θα ήταν, μέσω τροπολογιών, να συμπεριλάβουμε και άλλο σημείο. Να ζητήσουμε από τον Σέρβο, τον Πρωθυπουργό που επισκέφτηκε το Κωσυφοπέδιο την περασμένη εβδομάδα, ότι όταν επισκέφτεται τι σερβικέ κοινότητε στο Κωσυφοπέδιο, που είναι σημαντικό, να προγραμματίζει και επισκέψεις με τον Πρωθυπουργό του Κωσυφοπεδίου. Ε, είναι στοιχειώδες αυτό για τις καλές ε, σχέσεις. Πρέπει να συναντάς τον ομόλογό σου στη χώρα που επισκέπτεσαι. Πέραν αυτού, καλώς αναφέρεις τις εκλογές για τα Συμβούλια των Εθνικών Μειονοτήτων που έγιναν εκλογές τον Οκτώβριο του 2014. Υπάρχουν πολλοί Ρωμά ε, που είναι ανάμεσα στους Σέρβους και ζητούν άσυλο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σερβικές αρχές πρέπει να κινηθούν ε, ούτω ώστε να διευκολυνθεί η ένταξη των Ρωμά στην κοινωνία της σερβική. Θα παρακαλούσαν λοιπόν να φυγούν και αυτά. Και κατόπιν συζητήσεων του τους Είναι σαφές αυτό που είπατε ότι η επισημοποίηση των σχέσεων Κωσυφοπεδίου-Σερβίας είναι προϋπόθεση για την ένταξη της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να μεταρρυθμίσει δόντως και το σύνταγμά της η Σερβία. Αλλιώς δεν θα γίνει δεκτή η Σερβία. Εγώ υποστηρίζω την ένταξη της Σερβίας υπό αυτούς τους όρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτός μικροφώνου και ο Μπροκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή τον κύριο Μακάλιστερ που έξοχη έκθεσή του. Έχω μια ερώτηση όμως. Να θέσω ευθέω. Καλό θα είναι οι δυσκολίες να μεταφράζονται σε ευκαιρίες. Από τις 15 Ιανουαρίου η Σερβία ανέλαβε την Προεδρία του ΟΑΣΕ. Μήπως θα πρέπει λόγω παραδοσιακών σχέσεων με τη Ρωσία και εν ώψη της ευρωπαϊκής προοπτικής της Σερβίας που αναφέρεται και στην έκθεση μήπως θα ήταν καλό λοιπόν να συμπεριληφθεί σαν διαμεσολαβητή στην κρίση στην Ουκρανία το λέω αυτό διότι έχει μια θέση ουδέτερη. Και συμφωνώ με την ελευθεροτυπία που ανέφεραν οι συνάδελφοι να ενθαρρυνθεί η κυβέρνηση σερβική να κάνει όλα τα θαραλέα βήματα που χρειάζονται σε αυτή την κατεύθυνση. Και όπως έλεγε και η συνάδελφος η κυρία Λούνατσεκ, θα θέλαμε να δούμε μεγαλύτερη εμβάθυνση στα θέματα του περιβάλλοντος πολύ συχνά είναι τα πιο ακαθόδη προβλήματα των Δυτικών Βαλκανίων εν ώψη της μελλοντικής προσχωρήσεως των χωρών της ε, περιοχής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Oui, merci. Merci, Président. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να πω και εγώ πόσο εύστοχα τα λέει στην εκθεσή του ο Ντέιβιτ Μεκάλιστερ. Και θέλω να τονίσω δύο τινά. Πρώτα πρώτα το σημείο υπαριθμών 8 που αφορά τις κυρώσεις. Να τοποθετηθεί δηλαδή από αυτού η Σερβία. Και εμείς επίσης να αναρωτηθούμε αυτές οι κυρώσεις τι νομική βάση έχουν σε σχέση με το διεθνές δίκαιο. Δεν ξέρω ούτε καν κατά πόσο είναι νόμιμες τέτοιες κυρώσεις, αν προβλέπετε τέτοια διαδικασία. Πού στηρίζονται επομένω. Κάποιο άλλο τώρα το σημείο, η παράγραφος 23, εκεί που λέει για κάποια αναδιάρθρωση όσον αφορά τον κλάδο του φυσικού αερίου και του παρόχου. Ε, νομίζω ότι στη Σερβία αυτό δεν γίνεται. Αλλά και από τεχνικής πλευράς. Νομίζω ότι αυτό θα δημιουργήσει μια αβεβαιότητα, ανασφάλεια ενεργειακή στη χώρα. Πριν και εγώ πρόεδρε, και πρώτα να σας πω δύο λόγια για τη Σερβία. Πρώτα πρώτα κάτι διευκρινιστικό για την Βοσνία Ζεγοβίνη με τον οποίο και ασχολούμαι. Δεν το έχουμε αυτό στην μερσία διάταξη. Αλλά αναρωτιούνται γιατί δεν ασχολούμαστε με τη χώρα. Μα θα ασχοληθούμε την επόμενο μήνα θα γίνει αυτό. Οπότε και έτσι θα δοθεί η ευκαιρία στις καινούργιες αρχές της χώρας να ακούσουν τη γνώμη μας. Για τη Σερβία πάντως και την σχετική έκθεση γιατί στον κύριο Μακάλιστο και συμφωνώ μαζί του για το κεφάλαιο 23 και το κεφάλαιο 24 που θα πρέπει να να τα συζητούμε όσο γίνεται πιο σύντομα. Επίσης εκφράζω την έκπληξή μου γιατί ο Πρωθυπουργός Βούτζης είπε ότι, θα, ότι, ότι, ότι, ότι πληρώνονται οι μη κοινωνικέ οργανώσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να τον επικρίνουν. Αυτό δείχνει έλλειψη εμπιστοσύνη. Δεν μα πάει προ τη σωστή κατεύθυνση. Στο μέλλον να αποφεύγουν τέτοια πράγματα. Επίσης, Παραπέμπω στα είχε πει ο Επίτροπο Χάν τον ε, Δεκέμβριο για την σύγκληση των θέσεων. Όσον αφορά την Ρωσία. Έχουμε αυτό το παράδοξο σε σχέση με την Σερβία. να το βλέπουμε εμείς. Έχουμε το 52% που είναι υπέρ των σχέσεων με τη Ρωσία των στενότερων και επίσης έχουμε το 32% και στη χώρα που επίσης είναι ε, κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε η κυβέρνηση τώρα αποστασιοποιείται όσον αφορά την ε, ε, αντιπολίτευση, οπότε θα πρέπει και αυτό να το εξετάσουμε σε αυτή την οπτική γωνία. Για το 2011, επίσης να δούμε το τι έχει κάνει θετικά βήματα η Σερβία για τις τοπικές περιφερειακές πρωτοβουλίες. 17 όσον αφορά την βιωσιμότητα του κρατικού ε, ραδιοφώνου για τις ε, μειονοτικές γλώσσες για το 18 Επίση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι έχουμε κάποιο είδους καταγγελίες όσον αφορά την εκλογή των συμβουλίων για τις ε, εθνικές μειονότητες. Συγκεκριμένα που πρέπει τον χρόνο αγορευση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρόοδος ε, τη Σερβία σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό δρόμο είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί πρόκειται για μια χώρα με μια ιδιαίτερη ευθύνη και σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μεταξύ των χωρών στα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά και για τις υποψήφιες χώρες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σαφής η πρόοδος. Ο Ντέβιτ Μακάλιστερ τα ανέφερε αυτά εκτεταμένα. Αλλά αυτό που παραμένει ως υποχρέωση είναι το εξής. Η Σερβία, πέρα από τις δηλώσεις, θα πρέπει να ταχθεί υπέρ της προστασίας των εθνοτικών μειονοτήτων σε ό,τι αφορά και το δικαίωμα άσκησης της γλώσσας των μειονοτήτων. Εκτός αυτού, η σερβική κυβέρνηση θα πρέπει να κληθεί να προσαρμόσει τη σχετική νομοθεσία προκειμένου να μην γίνονται αποδεκτές ε, ομιλίες που καλούν στο μίσος σε ό,τι αφορά στη δήλωση της ΕΣΕΤ, ο κύριος Τάτσιτς δυστυχώς δεν θεώρησε ότι η κυβέρνηση στη Σερβία αντέδρασε όπως άρμοζε στις δηλώσεις αυτές. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ε, διαμόρφωση φυσιολογικών σχέσεων με τις γειτονικέ χώρες και επίσης να προσαρμοστεί η πολιτική και να συντονιστεί η εξωτερική πολιτική σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο διάλογο με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρειάζεται να διευκρινίσουμε πόσο σημαντικό είναι και σε ό,τι αφορά και τον διάλογο με τι γειτονικέ χώρε. Σε ό,τι αφορά τον ΟΑΣΕ, ενδεχομένω αυτό να σηματοδοτήσει μια εποχή εσωτερικών αλλαγών στην ίδια τη Σερβία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, κύριε Πετήρ. Δυστυχώ, Εξ όσων ε, καταλαβαίνω η έκθεση προόδου και το σχέδιο ψηφίσματος του κ. Μακάλιστερ δεν ε, εξετάζουν θέματα παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή παραβιάσεων του κράτους δικαίου σε περιπτώσεις ε, εγκλημάτων πολέμου. Από το 2010 η Σερβία σε νομοθεσία για την ε, δίωξη ε, εγκληματιών πολέμου στην Κροατία. Αυτό δεν σέβεται την επικυριαρχία της Κροατίας. Ο Μέλκο ε, Κροάτης πολίτης, κατηγορείται για εγκλήματα επικροατικής επικράτειας κατά ενός άλλου Κροάτη. Αν το ανοιχτούμε αυτό, δηλαδή θα μπορούσαν οι πολίτες ε, από τη Γερμανία, από την Αυστρία, από το Ηνωμένο Βασίλειο να περιληφθούν όλες ε, οι χώρες που προασπίστηκαν την ε, Κροατία θα μπορούσαν να βρουν στην ίδια μοίρα. Υπάρχει λοιπόν παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό το είδα μόνιμο όταν επισκέφθηκα τη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι χρειάζονται μεγάλε μεταρρυθμίσεις σε ό,τι αφορά την τήρηση του κράτου δικαίου. Και ότι πρέπει να τηρούνται οι κανόνε για του εγκληματίε πολέμου. Ζητούμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τα κεφάλαια και την πραγμάτευση με την Σερβία η τηρήση των ανθρωπινών δικαιωμάτων και σε ό,τι αφορά το Μάλιτς θεωρώ ότι να κοιτάξουμε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα συγχαρητήρια στον εισηγητή για αυτή την τόσο καλή ε, έκθεση για την πρόοδο της χώρας. Τελικά για τις μεταρρυθμίσεις είναι μεγάλη υπόθεση η πορεία προς ε, ένταξη. Για όλες τις χώρες που παίρνουν από τα μετασχηματισμούς και η Σερβία δεν θα ήταν εξαίρεση κοινωνική πολιτική, οικονομική πολιτική, πολιτικέ μεταρρυθμίσει έχουν ακόμα δρόμο μπροστά του, βέβαια σε και ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όλο ένα και περισσότερε δράσει αναλαμβάνει ώστε να υπάρχει μια κοινή, το τονίζω κοινή πολιτική ασφάλεια και εξωτερική πολιτική οπότε θα δίνεται ευκαιρία στη χώρα να προοδεύσει και άρα δεν θα πρέπει να αντιδρά σε μια ε, συνεπή ε, προσέγγιση προς την Ρωσία σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να επιδείξει η χώρα αλληλεγγύη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Θα έπρεπε να είναι πιο κοντά στις ε, ενωσιακές απόψεις για αυτή την πολιτική και ελπίζω ότι τα μέσα επόμενα χρόνια να δούμε μια πιο συνεπή γραμμή της Σερβίας σε σχέση με αυτό το θέμα. Πάντως, μόλις παγιωθούν οι τακτικές διαπραγμάτευσεις με την Ρωσία, θα έχουμε κάποια κεφάλαια τα οποία πλευρά Σερβίας θα είναι πιο προχωρημένα και θα πρέπει όλοι. αυτά να ανοίξουν όσο γίνεται πιο νωρίς και επίσης η Σερβία να συμμορφωθεί όπου πρέπει για μην αναβάλει. Ελπίζω ότι αυτό το σχεδιογημένο θα αποτελέσει μια στέρεη βάση για να προχωρήσουμε. Thank you, Chairman. I'm... Επόμενος. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που όλοι αυτοί οι είπαν τόσα πολλά για τις θέσεις της Σερβίας σε σχέση με τον ΟΑΣΕ. Η κυρία Μογκερίνη την περσμένη εβδομάδα μας μίλησε ότι θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι μια υπερδύναμη ειρήνης Έχουμε βέβαια τι σχέσεις σχέσει Σερβία και Ρωσία. Να, τώρα η ευκαιρία, που κάτι το οποίο είναι υπέρ τη ασφάλεια στην περιφέρεια, να δούμε την μοναδική αυτή θέση τη ε, Σερβία. Και αυτό το αναφέρει ο κ. Μακάλιστερ. Και ότι θα πρέπει να έχουμε κάποια ευθυγράμμιση στην εξωτερική πολιτική με την ε, Ρωσία. Άκουσα και την κυρία Λούνατσεκ Συμφωνώ κύριε Λούνατσικ και όσοι ίδιες θέσεις έχω όσον αφορά τους τσιγκάνους και τα προβλήματα σε πολλές χώρες. Μίλησε ο κρότης συνάδελφος και όλοι μας θέλουμε τελικά η Σερβία να δεις προσπάθειες να ευοδοθούν. Και τότε θα πρέπει να δούμε ότι θα βρούμε τη πλήρω νομοθεσία σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη. Και τότε θα πάρα πολλέ εκκρεμίε υποθέσει θα τακτοποιηθούν και επίση τελικά αυτό θα φέρει και την συμφιλίωση των παλαιών εχθρών. Ευχαριστώ. Ευπρόσδεκτη έκθεση του κ. Μακάλιστερ. Χαιρετίζω τις προσπάθειες που έκανε. Σίγουρα έχει προχωρήσει η Σερβία, είναι αδιαμφισβήτητο. Έχω κάποια ζητήματα που θέλω να θίξω όμως. Οι σχέσεις με τη Ρωσία είναι ένα θέμα. Αναφέρθηκε και την προηγούμενη φορά. Ο κ. Μακάλιστερ κάλεσε την Σερβία να εξομαλύνει την εξωτερική της πολιτική, μάλλον να την συντονίσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι πολύ φιλικές σχέσεις με τη Ρωσία δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Τώρα, όσον αφορά την επικοδομητική πολιτική γειτονία, ξέρουμε ότι εκεί παραμένουν κάποιες εκκρεμότητες και θα πρέπει να τις κουβεντιάσουμε. Παραδείγματος χάρη, τα σύνορα του Δούναβη μεταξύ Κροατία Κροατίας και Σερβίας και διάφοροι, ε, διάφοροι εξαφανιστέντες, δεν ξέρουμε αγνοούμενοι που υπάρχουν ε, υπάρχουν και θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς που πρέπει να διαθετηθούν. Μετά το άνοιγμα των αρχείων των Ιουγκοσλαβικών. Δεν θέλουν οι σερβικές αρχές για την ώρα να το κουβεντιάσουν αυτό. Ο κύριος Μάριτς και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ένα άλλο θέμα και η δικαιοδοσία της Σερβίας όσον αφορά ε, τα εγκλήματα πολέμου που πρέπει να εξεταστεί. Οι εθνικές μειονότητες μετά αναφέρεται η αμοιβαιότητα που είχε συμφωνηθεί αυτή πριν το 2005, η αμοιβαιότητα μεταξύ Κροατίας και Σερβίας. Οι Σέρβοι στην Κροατία έχουν τρει έδρε στο Κοινοβούλιο, ενώ οι Κροάτε, που είναι η τέταρτη μειονότητα στη Σερβία, δεν έχουν καμία τέτοια εγγύηση. Άρα και αυτό θα πρέπει να αναφέρεται στο μέλλον. Και το θέμα των ομιλιών μυσαλλοδοξία ε, για τον Σέσελ που είναι και κλιματίας πολέμου. Αυτές, αυτοί οι λόγοι πρέπει να ακούγονται σήμερα. Αλλά δεν έχουμε ακούσει κάποια καταδίκη εκ μέρου των σερβικών αρχών όσον αφορά τι ομιλίε μυσαλλοδοξία. Ακόμα διαμορφώνεται η έκθεση, άρα υπάρχουν περιθώρια για κάποιε βελτιώσει με την πάροδο του χρόνου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο Μακάλιστερ για το σχέδιο ψηφίσματο για την έκθεση πρόοδου για τη Σερβία. Καλό θα ήταν για όλη την ε, περιοχή και για την ενίσχυση της δημοκρατίας αν η πορεία της Σερβίας ε, κινούταν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και από νομικής άποψης. Ε, να τονίσω κάποια στοιχεία τα οποία θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά στην έκθεση αυτή. Εδώ στην αίθουσα αυτή Είχαμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Κριτάτσι πριν από 1,5 μήνα. Και πριν από ένα 1,5 μήνα από σερβικής πλευράς, από τον κύριο Πούτσης και τον κύριο ε, Νίκολιτς που ήταν μαζί στο ίδιο κόμμα με τον κύριο Σέσσερ πριν από κάποιο καιρό συζητήσαμε το θέμα των ε, ομιλιών μη και τη ρητορία πολέμου του ΣΕΣΕΛ. Βλέπουμε ότι αυτή η ρητορική υπάρχει ακόμα στα μέσα ενημέρωση. Δεν είναι, θεωρούμε, θετικό ε, μια χώρα που βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην τηρεί τέτοια πρότυπα για τα έγκληματα πολέμου. Κατά δεύτερον, ένας νόμος όπου η Σερβία θέλει σε ό,τι αφορά το ΣΕΣΕΛΕ το δικαστήριο της Χάγης. Το άρθρο 3 σε ό,τι αφορά τα εγκλήματα πολέμου αναφέρει ότι θέλει καθολική ε, δικαιοδοσία η Σερβία για τα εγκλήματα πολέμου. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει αυτό σε ό,τι παραμελικούλα. Έτσι, συμφωνώ με του ε, συναδέλφου σε ό,τι αφορά την εξωτερική της πολιτική. Θα πρέπει να αποφασίσει προς τα πού θέλει να κινηθεί η Σερβία αν θέλει να κινηθεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να υπαχθεί στη γενικότερη εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πόσο μάλλον που κατέχει, και την Προεδρία του ΟΑΣΕ. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин σας ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Θα συμφωνήσω με τις ευχαριστίες προς τον εισηγητή και εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ αξιο πρέπει οι προσπάθειες που έκανα. Αλλά συμφωνώ και καταλαβαίνω και τα θέματα των Κροατών συναδέλφων. Θεωρώ ότι αυτά συνδέονται και με την ελευθερία έκφραση. Υπάρχουν προβλήματα και σε ό,τι αφορά τι εθνικέ μειονότητε. Να σα επιστήσω την προσοχή και σε ένα πρόβλημα το οποίο έχει να κάνει με την τρική γλώσσα στο Μπουζίλικραντ και στις γειτονικέ περιοχές. Πάντα υπάρχουν λοιπόν δικαστικέ αγωγές κατά των ηγετών αστυνοτικών μειονοτήτων όπως τον Δημήτρη Δημήτροφ, Μοζίλικρατ, συγκεκριμένα παραδείγματα σας αναφέρω, αλλά και κατά δασκάλων. Μπορώ να σας αναφέρω ονόματα δασκάλων στους οποίους στερείται το δικαίωμα να διδάξουν επειδή διδάσκουν στη μητρική τους γλώσσα. Αυτά είναι προβλήματα στο σερβικό κράτος και θα πρέπει να λεφθούν υπόψη να αντιμετωπιστούν. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη μελλοντική ενδεχόμενη προσάρτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να αποφασίσει Ποια θα είναι η μελλοντική της πορεία η Σερβία. Επενώ το έργο του εισηγητού, την ενέργεια που διέθεσε για την όλη διαδικασία. Χαίρομαι επίσης διότι η έκθεση είναι ισορροπημένη, εμπεριέχει τα βασικά πολιτικά στοιχεία, τα θέματα, ερωτηματικά αλλά και επιτεύγματα. Κατά την άποψή μου χρειάζεται υποστήριξη και βοήθεια για τη Σερβία και τη σερβική κυβέρνηση, ούτως ώστε να μπορέσει να προχωρήσει με το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Χρειάζεται κατά την άποψή μου να μπουν και άλλες παρατηρήσεις στην έκθεση, όπως για το θέμα των Εθνικών Συμβουλίων και των Εθνικών Μειονοτήτων. Ποια είναι τα δικαιώματά τους, ε, πώς εφαρμόζονται αυτά τα μέτρα ή τα συμβούλια και εν ώψη του σχεδίου δράσεως για το κεφάλαιο 23 που διαμορφώνεται από τη σερβική κυβέρνηση κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά είναι τα σημεία που θα ήθελα να αναφέρω σε αυτές τις σύντομες παρατηρήσεις. Για μία ακόμη φορά ευχαριστώ τον εισηγητή για την καλή δουλειά που έκανε. Ευχαριστώ. Thank you very much, uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Μακάλιστερ, αξιότιμα μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται τη γενική αξιολόγηση του εισηγητού και νομίζω ότι το ψήφισμα καλύπτει σωστά την πρόοδο που επετέφθη στη Σερβία το 2014. Παραμένει η Σερβία αφοσιωμένη στο πρόγραμμά της για Ευρωπαϊκή Ένωση και στις μεταρρυθμίσεις της και η Σερβία έπαιξε θετικότατο ρόλο στο όλο περιφερειακό πλαίσιο. Το ψήφισμα στηρίζει τις συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις στη Σερβία, όπως οικονομικό τομέα, στον οικονομικό, τον κοινωνικό τομέα και υπογραμμίζει σαφέστατα τις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πολλές ανησυχίες ακούστηκαν και τώρα στη συζήτηση. Σημειώνω ιδιαίτερα την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, την ελευθερία της έκφρασης και την ευθυγράμμιση με την κοινή εξωτερική πολιτική. Είναι ανησυχίες που ενστερνίζεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ενταξιακέ διαπραγματεύσει με τη Σερβία ξεκίνησαν εδώ και ένα χρόνο, 21 Ιανουαρίου του 2014. Συνεχίζεται ως προγραμματίσει η διαδικασία, θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο φέτος. Μαζί με τον εισηγητή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιμένει το άνοιγμα των πρώτων κεφαλαίων. Αυτό εξαρτάται κατά πολύ από τη δυνατότητα της Σερβίας ποιοτικά να πετύχει αποτελέσματα, ποιοτικά αποτελέσματα για το κράτο δικαίου και για την εξομάλυνση των σχέσεων με το κοσυφοπέδιο. Βασικοί τομείς. Πρέπει γρήγορα να συζητηθούν στην ενταξιακή διαπραγματεύση. Στη διαμόρφωση του διαπραγματευτικού πλαισίου. Σε όλους αυτούς τους τομείς θα στηρίξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη Σερβία. Με το ίδιο πνεύμα και την ίδια ένταση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ο πρόεδρος συνεχίζει εκτός μικροφώνου, δεν τον ακούνε οι Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι και συνάδελφοι, πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω τον κύριο Κούκαν, τον Σκιώδη εισηγητή, και τους άλλους συναδέλφους, γιατί ήταν η συμβολή τους πολύτιμη. Και προσωπικά θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολλά κοινά σημεία και αυτή η, αυτό το κείμενο, αυτό το ψήφισμα στον Μάρτιο στην Ολομέλεια θα περάσει με μια ευρία πλειοψηφία. Τώρα να μην επισέλθω στι λεπτομέρειε γιατί πιέζει ο χρόνο. Όμω να σα πω κάποιε παρατηρήσει παρατηρήσεις πρώτα-πρώτα όσον αφορά την εξωτερική πολιτική. Κύριε Καστάλντο, τόνισα ότι θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θετικό το θα ασκήσει το 2015 η Σερβία την Προεδρία του ΟΑΣΕ και επίση τόνισα ότι θα μπορούσε ε, αυτός ο ρόλος να χρησιμοποιεί και σε σχέση με αναζήτηση λύσεων όσον αφορά το πρόβλημα ε, Ρωσίας-Ουκρανίας. Πάντως, αν θέλουμε μια υποψήφια χώρα να ευθυγραμμίζεται πλήρως, αυτό αφορά και την εξωτερική πολιτική. Και όσον αφορά την κατάσταση σε Ρωσία και Ουκρανία, υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ ημών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σερβίας. Γιατί η Σερβία ήταν υπέρ της ε, αντοχής ακρότητας της ε, Ουκρανίας αλλά δεν προσπέραψε το ψήφισμα του ΟΗΕ το σχετικό και σε σχέση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου για τα εμπάργου και για τα άλλα μέτρα κατά της ε, Ρωσίας όσον αφορά την παράνομη κατοχή της Κρυμαίας ούτε τότε συντονίστηκε. Τώρα όσον αφορά τα ενεργειακά στην έκθεσή μου εγώ τόνισα ότι σημειώθηκε πρόοδος στον ενεργειακό τομέα και ιδίω όσον αφορά τον ηλεκτρισμό, τα ανανεώσιμα, ε, την αποτελεσματική χρήση ενέργειας όμως χρειάζεται να προσπαθήσει περισσότερο η χώρα ούτω ώστε ε, να ρυθμιστεί το θέμα της τιμολογικής πολιτικής για ε, τον ηλεκτρισμό και επίσης και για το φυσικό αέριο. Συμφωνώ με την κυρία Λούνα ότι η Σερβία θα πρέπει να καταβάλει πιο σημαντικές προτάσεις πρόσεχε προσπάθειες για να μπορέσει να φτάσει στους στόχους που έχει τάξει. Τώρα το τελευταίο που θα σα αναφέρω είναι κάτι το οποίο ε, διάβασα στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων yes, χθες, ε, και το DPA, το πρακτορείο είπε ότι η Σερβία απείλησε ότι στις 9 Δευτέρου ε, θα δυναμητήσει τον διάλογο εάν το κοσμοπέδιο αποφασίσει να καταλάβει ε, το ορυχείο μεταλλείο στην Τρέψα το θέμα είναι περίπλοκο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτού του είδους ο διάλογος της 9 Φεβρουαρίου να γίνει ο διάλογος υψηλού επίπεδου και έτσι να έχουμε πρόοδο, να έχουμε περισσότερη εξομάλυνση στις σχέσεις Βελιγραδίου Πρίστινα. Οπότε γι' αυτό και ελπίζω ότι αυτά που είπε το Γερμανικό Προεκτροειδήσεων ή δεν είναι ανακριβή ή δεν θα συμβούν. Ευχαριστώ όλους και ειδικά τους ε, σχεδοσυγητές και υποβάλλεται ε, τροπολογία μέχρι τι 27 Ιανουαρίου το μεσημέρι. Jerry Cooper is around the corner. As I followed this debate just now, I was reminded is the... Και η συζήτηση, λέει ο Πρόεδρος. Μου κάτι μου θύμισε τώρα. Είναι εδώ ο κύριος λέει. Όλα αυτά που λέγαμε για την Σλοβενία. Αυτά θυμήθηκα. δεν μπορεί παρά να έχουμε καλή πίστη και θετική αντιμετώπιση, αλλιώς θα τα βρούμε μπαστούνια. Και τώρα κύριε Λόντσα και για το Κασικοπέδιο. Ευχαριστώ πρόεδρε, συνάδελφοι. Το θέμα είναι, η διεύρυνση και η έκθεση διεύρυνση και πρόοδου για το κοσυφοπέδιο και η δική μου η έκθεση γι' αυτό. Στην έκθεση μου αναφέρω ότι υπήρξε σημαντική πρόοδο στο τελευταίο χρόνο, από την τελευταία έκταση που έγινε, σε ό,τι αφορά τις εκλογικές διαδικασίες, ότι οι εκλογές ε, το Μάιο και τον Ιούνιο του 2014 διοργανώθηκαν με σωστό τρόπο και ότι υπήρξε συνέχεια μετά τις δημοτικές εκλογές του προηγούμενου έξαμην. Ήταν πολύ καλά τα πρότυπα, πολύ καλός ο τρόπος διεξαγωγής εκλογών στο Κωσυφοπαίδιο. Παρ' όλα αυτά, τονίζω ότι υπήρξε πολιτικό τέλμα επί έξι μήνες και τώρα καλωσορίζει το γεγονός ότι μετά αυτή την περίοδο σχηματίστηκε κυβέρνηση. Είχα την ευκαιρία να είμαι εκεί όταν τελικά σχηματίστηκε η κυβέρνηση και η νέα κυβέρνηση λοιπόν θα πρέπει να ε, δώσει συγκεκριμένα αποτελέσματα στους πολιτιστικούς υποπεδίους, την καταπολέμηση της διαφθοράς, τη βελτίωση της οικονομικής ε, και κοινωνική κατάσταση των πολιτών. Ελπίζω λοιπόν να κάνει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις με τόλμη και θάρρος η κυβέρνηση. Δύο θέματα έχω να σχολιάσω αρνητικά σε ό,τι αφορά το σχηματισμό τη νέα κυβέρνηση, Δύο μόνο γυναίκες μεταξύ 21 υπουργών και συνομίλησα με κάποιους εκπροσώπους. Υπάρχουν τουλάχιστον στο Κοινοβούλιο κάποιες γυναίκες πρόεδροι ε, κοινοβουλευτικών επιτροπών, αλλά και εδώ χρειάζεται αύξηση. Και επίσης ανησυχία για ε, τον διορισμό ατόμων επί των οποίων δεν υπάρχει συνένεση αμφιλεγόμενων προσωπικότητων. Αυτό αξίζει να το αναφέρουμε. Αυτά για το σχηματισμό της κυβέρνησης. Φυσικά, όπως είπα, η σημασία της πραγματικής βελτίωσης της οικονομικής και της κοινωνικής κατάστασης είναι θέματα κλειδιά και επίσης αναφέρθηκα στο ότι υπάρχει πρόοδο σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση του δικαστικού σώματος και από κοινού με τη Ulex αναφέρθηκα στις κατηγορίες διαφθοράς κατά της Γιούλεξ που βγήκαν στο προσκήνιο στο τέλη του 2014. Ξέρουμε ότι είναι σημαντικό αυτές οι κατηγορίες να αντιμετωπιστούν με γρήγορο τρόπο. Καλωσορίζω και την ταχεία αντίδραση της κυρίας Μογκερίνη που πολύ γρήγορα αποφάσισε να διορίσει ειδικό αντιταλμένο για την εξέταση του θέματος αυτού. Για το σύνολο του δικαστικού σώματος και για την συνέλευση του κοσυφοπεδίου ζητούμε να περάσει νομοσχέδιο για να υπάρξει λειτουργικό τέτοιο σώμα. Χαίρομαι που τον Αύγουστο του 2014 έγινε μια πρώτη έξεση, ότι υπήρχε μια συμφωνία με την κυβέρνηση των κάτω χωρών να υπάρξει για το ειδικό δικαστήριο συνεργασία και ελπίζουμε λοιπόν το πακέτο αυτό να περάσει από την Εθνοσυνέλευση των Συντήματων Τώρα, σε ό,τι αφορά άλλα θέματα η εκκίνηση του, της Συμφωνίας και Σύνδεσης τον Ιούλιο του 2014. Πολύ θετικό. Ελπίζω το Συμβούλιο, και εδώ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση, να εγκρίνει το συντομότερο δυνατόν τη συμφωνία αυτή, προκειμένου το 25 να μπορέσει να συμμετάσχει σε όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Άλλε πτυχέ είναι σαφές ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να συνεχίσει και θα πρέπει να βελτιώσει την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος σε όλα τα επίπεδα. Γιατί εξω όσων γνωρίζουμε και όπως γνωρίζουμε και από άλλες χώρες, όχι μόνο το κοσμοπεδίο, η διαφθορά αποτελεί εμπόδιο στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και στη δημοκρατική άλλωστε ανάπτυξη. Άλλα ζητήματα που μας ανησυχούν για το κόσμο στο κοσμοπεδίο είναι ο χάρτης πορείας για την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Σημαντική πρόοδος έχει γίνει από την πλευρά της κυβέρνησης. Τέσσερα νομοσχέδια λείπουν και όλοι από πλευρά της κυβέρνησης με διαβεβαιώνουν ότι θα προσπαθήσουν να τα ολοκληρώσουν το δυνατόν. Δυστυχώς επίσης είναι μεγάλος ο αριθμός ε, που, των πολιτών από το πέδιο που έφυγαν από το Κωσυφοπέδιο για τη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, Ρώμα, Σκάλι αλλά και ε, Αλβανή. Θα πρέπει η κυβέρνηση του Κοσμοπεδίου να δώσει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στον κόσμο αυτό. Θα ήθελα να επίσης να ξεκαθαρίσω προς τους πρωθυπουργούς και τους υπουργούς εσωτερικών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι και πάλι το Κωσυφοπέδιο είναι η μοναδική χώρα της περιοχής όπου οι πολίτες δεν έχουν δικαίωμα ελεύθερα να ταξιδεύουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι θα πρέπει να γίνει λοιπόν αυτό. Ένα άλλο θέμα στο τέλμα στο σχηματισμό της κυβέρνησης ήταν και η έλλειψη επενδύσεων στη χώρα των τελευταίων εξάμεινων. Και λοιπόν για το θέμα αυτό χαίρομαι που σχηματίστηκε η κυβέρνηση. Ελπίζω οι επενδύσεις να ξεκινήσουν και πάλι σε ό,τι αφορά το διάλογο μεταξύ της Σερβίας και του Κωσυφοπεδίου, ο οποίος ήδη αναφέρθηκε στην προηγούμενη συζήτηση, δυστυχώς λόγω των συνθήκων και στις δύο χώρες η όλη διαδικασία έχει επιβραδυνθεί. Και δυστυχώς επίσης η συμφωνία του Απριλίου δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα πλήρως και καλό και τις δύο χώρες να προχωρήσουν. Επίσης ε, με λυπή ένα στοιχείο της συμφωνίας που δεν έχει εφαρμοστεί, ναι. αν και δεν είναι το μόνο, είναι η έλλειψη των διεθνών κλήσεων. Αν θέλει κανείς να πάρει τηλέφωνο κάποιος στο κοσμοπέδιο, ακόμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κωδικό Σλοβενίας ή Μονακό. Αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ναι. Είναι σημαντικό, θεωρώ. Και η εκλογές για δημάρχους στο βόρειο τμήμα του έλαβαν χώρα. Ελπίζω να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύντομα. Ένα τελευταίο θέμα τώρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει η Ρώμα, η Ασκάλη και οι Αιγύπτη να ανταχθούν καλύτερα σε ό,τι αφορά το σεβασμό των δικαιωμάτων. ένα στατικό Σημάδα ήταν ε, η διοργάνωση του Gay Pride πέρσι. Εντυπωσιακό ο αριθμό των συμμετεχόντων και η κυβέρνηση έχει ένα σχέδιο για την κοινότητα των ΛΟΑΔ στη χώρα. Προσβλέπω λοιπόν στην καλή συνεργασία με τους κοιότες και ελπίζω ότι... Α, συγγνώμη, ξέχασα ένα θετικό στοιχείο σε ό,τι αφορά τη διεθνή αναγνώριση του πεδίου. Η πλήρης αναγνώριση της Ολυμπιακής Επιτροπής ε, στην Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Αυτό τι σημαίνει ότι οι αθλητές ε, του κοσμοπεδίου θα μπορέσουν να συμμετέχουν με τα ονόματά τους, με τη σημαία τους στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σημαντική πρόοδος. Θα πρέπει να είναι πλήρες αναγνωρισμένο μέλος ε, στον ΟΗΕ το κοσυφοπαίδιο, αλλά και στη Europol και στην Interpol για την καταπολέμηση του εγκλήματος. Και να κλείσω με ένα σχόλιο το οποίο επαναλαμβάνω από το 2010 ότι καλό και τα πέντε κάτι μέλη που δεν έχουν αναγνωρίσει το κοσμοπέδιο να το πράξουν γιατί είναι απλά γεγονός και θα βοηθούσε και τα ευρωπαϊκά προγράμματα αν συμμετείχαν και τα 28 κράτη-μέλη σε αυτό το όραμα του κοσμοπεδίου. Ευχαριστώ. Euh, Ευχαριστώ απείρως κύριε Πρόεδρε. Έχω τρία σχόλια σαν αφορά την έκθεση της κυρίας Λούνατσεκ, συγχαίροντας την για τη δουλειά που έκανε. Πρώτη παρατήρηση, το θέμα που αναφέρθηκε, έκκληση προς τις πέντε χώρες που δεν αναγνώρισαν ε, το κοσυφοπέδιο είναι ένα θέμα που μας διαχωρίζει. Υπάρχουν πέντε χώρες κράτη-μέλη που δεν το έκαναν και το συζητήσαμε αυτό στο Κοινοβούλιο, πανηλημένα στην παράγραφο 12, η κυρία Λούνα Τσεκ συσχετίζει και στενά την αναγνώριση από τις πέντε χώρες με την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Πρίστινα και Βελιγραδίου. Δεν συμφωνώ η εξομάλυνση σχέσεων Πρίστινα Βελιγραδίου πρέπει να λάβει η χώρα εκτός των αποφάσεων των πέντε, των πέντε μελών που δεν έχουν αναγνωρίσει ακόμα το κοσυφοπέδιο ως κράτος. Νομίζω ότι η εξομάλυνση λοιπόν δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από τη στάση πέντε χωρών. Παράγραφος 15. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε ότι Θέλουμε η Εουλέξ να συμμετέχει περισσότερο στις όλες τις διαδικασίες και ότι υπάρχει σχέση μεταξύ δράσεως Εουλέξ και τοπικής αυτοδίκησης. Παράγραφος 18. Το θέμα διαλόγου Σερβίας Κωσυφοπεδίου πρέπει να είμαστε σαφέστατοι. Επί των γεγονότων είναι πολύ περίπλοκος ο διάλογος, οφείλεται όμως αυτό στην όλη καθυστέρηση από πλευράς ε, λόγω της συστάσεως των αρχών στην Πριστίνα. Θα πρέπει αυτό να το αναφέρουμε και ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ο κύριος Παντζέρη, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την συνέδριο Λούντζεκ. Πάνω από πέντε χρόνια παρακολουθώ αυτή την υπόθεση. Και υπάρχουν ακόμα και πάρα πολλές σκιές και εμβολίες που τις έχουμε διασκεδάσει. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει πώς θα προχωρήσει ο δημοκρατισμός της ε, χώρας, πώς επίσης θα προοδεύσει ο διάλογος Σερβίας και Κωσυφοπεδίου. Να βάλουμε υπόψη ότι μετά από έξι μήνες σχηματίστηκε η κυβέρνηση και θα πρέπει να πούμε δύο ότι αυτή η κυβέρνηση ότι θα πρέπει να δούμε για τη σύνθεση αυτής της κυβέρνησης. Δεν μπορούμε βέβαια να παρέμβουμε, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και φυσιολογικές προσωπικότητες. Ρεαλιστικά τα βλέπει η κυρία Λούνατσερ για το σχέδιο στο κοσυφοπαίδιο, αλλά θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, να μην δικαιολογούμε κάποιες καθυστερήσεις που σημειώνονται και θέλω να σταθώ στα εξή σημεία. Ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και των δικαστών κατά πολέμηση διαφθορά. Να δούμε το ότι έχουμε μόνο τυπική, ονομαστική πρόοδο κάποιου νόμου που περάσανε, αλλά τα πράγματα καθόλου δεν άλλαξαν. Έχουμε επίση σοβαρά εγκλήματα, τα οποία δεν έχουν διωχθεί και κυριαρχεί η παρανομία. Κάτι άλλο τώρα που θα πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερως, το ρόλο της Ιούλεξ. Πέραν των ερευνών για την διαφθορά, να δούμε για τον ρόλο της Ιούλεξ μετά από όλη αυτή τη χρονική διαδρομή. Ακόμα. Δεν έχει τονιστεί αρκετά το ότι συνεχίζει τη διαφθορά, ονομαστική ήταν μόνο η κάθραση, Οπότε τα έχουμε πει και ξαναπεί, αλλά θα πρέπει ίσω να έχουμε κάποιο είδους έλεγχο, να γίνει διαδικασία ελέγχου στην Γιούλεξ για να δούμε το πώς θα λειτουργεί όπως πρέπει. Τώρα για τι μεταρρυθμίσεις οικονομικές και κοινωνικέ. Δεν αρκεί το ότι μετά από έξι μήνες μετά από όσα η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο και επειδή έγινε η κυβέρνηση θα έχουμε επενδύσεις. Πρέπει να γίνουν σε βάθος μεταρρυθμίσεις. Αυτό να συζητήσουμε. Thank you very much, Mr. Chairman. Congratulations to... Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια στην κυρία στην κυρία Ουλρίκε. Ο Λούνατζεκ θα πει πολύ καιρό παρακολουθεί τα πράγματα, ε, έχει τη γνώση, την εμπειρογνωμοσύνη και αυτό τα μετέφερε στην έκθεση. Έχω μια-δυο παρατηρήσει όσον αφορά τι εκεί εξελίξει. Είναι θετικό ότι τελικά έχει κυβέρνηση η χώρα. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρουν και θα αντιμετωπίσουν όλες τις δυσκολίες. επιγόντως θα πρέπει η χώρα να πετύχει οικονομική ανάπτυξη. Έχουμε σε κάποιο κομμάτι του πληθυσμού πάνω από 40% ανεργία, χαμηλούς μισθούς και πλήστεται ιδιαίτερα η νεολαία. Θα πρέπει επομένω η καινούργια κυβέρνηση να δώσει κάποιε υψηλέ προτεραιότητε για κάποια ζητήματα, όπω καταπολέμηση διαφθορά οργανωμένου κλίματο παραμένει. Αυτό ένα από τα σπουδαία προβλήματα. Χρειάζεται επίση να υπάρξει ένα ειδικό δικαστήριο και είδατε τι είπε η ειδική task force στην έκθεσή τη. Επίση. σύμφωνα με την εισηγήτρια ότι θα πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία, η απορρίθμιση, η απελευθέρωση σχετικά με τις θεωρίες διαβατηρίων ξέρω ότι τώρα η συγκυρία είναι μάλλον αρνητική όσο εγκαταλείψουν τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά πάντως η τάση αυτή θα πρέπει να είναι και να συνεχιστεί αυτού του είδους η, χαλάρωση. Κάτι άλλο τώρα, το οποίο και αυτό δεν είναι τόσο δημοφιλές. Πρόκειται για τις κατηγορίες διαφορά στην Ulex. Αυτό θα πρέπει αποφασιστικά να το αντιμετωπίσουμε και με διαφάνεια. Να γίνει μια πλήρης έρευνα και αντιμετώπιση. Τώρα, για το διάλογο Βελιγραδίου και Πρίστινας. Θα πρέπει και οι δύο πλευρές να συνεχίσουν τις προσπαθίες τους, να έχουν καλοπιστία και νομίζω θα πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να υπάρχει η σωστή ατμόσφαιρα για τη συνέχιση της πορείας αυτής. Ευχαριστώ. Επόμενος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να επενέσω αυτή την πληρέστατη έκθεση της κυρίας Λούνατσεκ. Προσβλέπω σε περαιτέρω συνεργασία μαζί της με την πρόοδο της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τη χώρα που συζητούμε. Όσον αφορά την πρόοδο που έχει πετύχει το Κωσίφο λοιπόν, Έχουμε δύο βασικές παράμετρους που πρέπει να λάβουμε υπόψη για να δούμε τι πρόοδος έχει επιτευχθεί. Τι γίνεται με τη διαφθορά που είναι ευρέως δεδομένη και τι γίνεται με το κράτος δικαίου και την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Κάτι άλλο που θα επηρεάσει εξελίξεις είναι η υψηλή ανεργία που έχει ξεπεράσει το 50% κυρίως ανάμεσα στους νέους. Χρειάζεται μεγαλύτερη ενότητα και επικρατεί μια πόλωση για λόγους πολιτικούς. Σχηματίστηκε κυβέρνηση τελικά μετά από πολλά προβλήματα και αυτή, ο σχηματισμός κυβέρνησης δημιούργησε το χώρο ούτω ώστε να προθυθεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα στη χώρα. Ελπίζω αυτό να ισχύει. Αν γίνει οτιδήποτε διαφορετικό θα υπάρξει περαιτέρω διχασμός και θα πρέπει να υπάρχει προοπτική ευρωπαϊκή για την πολύ φτωχή αυτή χώρα όσον αφορά τις εικασίες και τις κατηγορίες, καταγγελίες για διαφθορά στην Ulex. Αυτό δημιουργεί ερωτηματικά όσον αφορά τους θεσμικούς φορείς Ευρωπαϊκής Ενώσεως που κινούνται σε ένα τέτοιο περιβάλλον όπου υπάρχουν καταδίκες ε, για λόγους πολιτικούς. Οι έρευνες που θα διεξαγάγει η κυρία Μογκερίνη. Ελπίζω να εξηχνιάσουν το θέμα και θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στι σχέσει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ενώση και Κωσυφοπεδίου. Θα ανοίξει ο δρόμο για το Κωσυφοπεδίο και θα συνεχιστεί και το έργο των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Φορέων. Ε, χωρίς τη βοήθεια αυτή δεν θα υπήρχε συμφωνία Κωσυφοπεδίου Πριστίνα και χωρίς τη συνεργασία θα είχαμε μεγαλύτερα προβλήματα όσον αφορά την σταθερότητα την περιφερειακή. Αυτά και ευχαριστώ. Itself, John Basky, Mr. John κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, ε, ήταν χωρίς μικρόφωνο, γι' αυτό η προφορά του ονόματος δεν ήταν τόσο καλή. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμε, Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, με την ιδιότητά μου ως εισηγητής ε, από το ECR θα πρέπει να πω ότι συμφωνώ με τη θετική αξιολόγηση σε ό,τι αφορά το κείμενο της κυρίας Λούνα Τσέκ. Έχω εντυπωσιαστεί ιδιαίτερος από την σοβαρή της στάση και από τη σκληρή δουλειά που έχει κάνει. Δεν είναι αυτονόητο να τονίζουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το κοσυφοπέδιο, η υψηλή ανεργία, το κάτω δικαίου, η καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσει το κοσυφοπέδιο το διάλογο με τη Σερβία σε ό,τι αφορά τα κοινά σύνορα. Αυτό που κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ ανησυχητικό είναι η αιτιάσεις για διαφθορά στην ε, Ulex. Ξέρετε ότι το έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό και καλέσαμε από τότε τον ε, αντιπρόσωπο να μας ε, αναφέρει ποια άτομα συγκεκριμένα θα πρέπει να δράσουν. Το μέλλον του κοσφοπεδίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται από το κατά πόσο οι σχέσεις μεταξύ Βελιγραδίου και Πριστίνα μπορούν να διαλευκαθούν. Επιτρέψτε μου, κυρία Λούνατσεκ, να σας συγχαρώ εκ νέου. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Eh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Βάτμαντ. Θα ήθελα και εγώ να ξεκινήσω χαίροντα την κυρία Λούνατσακ για την καλή έκθεση που έχουμε μπροστά μα σήμερα. Φυσικά είναι σημαντικό αν ω Ευρώπη θέλουμε να μιλήσουμε με μία φωνή. Είναι σημαντικό λοιπόν να αναγνωρίσουμε το κοσυφοπέδιο, την ανεξαρτησία του. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι γίνεται έκκληση στα πέντε κράτη που δεν έχουν ακόμα αναγνωρίσει το κοσυφοπέδιο να το πράξουν. Έχω κάποιες προσθήκες και κάποιες τροπολογίες να κάνω. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε για παράδειγμα να καλέσουμε το Κόσυφο παιδείο να επενδύσει στις ε, σχέσεις γειτονία με τις γειτονικέ χώρες. Ένα άλλο θέμα το οποίο επίσης δεν πρέπει να παραλείψουμε είναι ότι θα πρέπει να μιλήσουμε για την καλή ε, πολιτική για την ενέργεια. Έχουν προβλήματα βλέπουμε σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό και θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει σωστή ενεργειακή πολιτική προκειμένου να υπάρχει σωστή οικονομία. Τέτοια ζητήματα λοιπόν, μικροθέματα θα ήθελα να, περιλάβουμε, να συμπεριλάβουμε σε τροπολογίε, αλλά συνολικά θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω την κυρία Λούνατσεκ για την πολύ καλή προσέγγιση τη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ, την για το άριστο έργο της για αυτό το θέμα. Ενδελεχής και σε βάθος η δουλειά της και συμφωνώ με αυτά τα οποία ανέφερε για τη με το 4 και με το 5. Εκεί που αναγνωρίζεται το πρόβλημα της δικαιοσύνης, της καταπολέμησης, της διαφθοράς, ε, για κάποια βήματα για το ξύπνο χρήματος, αλλά Επίσης, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, θα πρέπει να τονίσουμε για το θέμα της τρομοκρατίας. Μέχρι πριν από λίγου μήνε, δεν είχε το Κόσοβο νόμο κατά τις δράσεις των τρομοκρατών και επίσης για των λεγόμενων ξένων μαχητών. Και υπήρχε το θέμα των εκλογών, οπότε δεν είχε περάσει ακόμα ο νόμο που έπρεπε και ε, πρόκειται για ένα πρόβλημα στη δικαιοσύνη που αφορούσε 43 πρόσωπα και μετά ε, είχαμε και πρόβλημα που αφορούσε υπόλοιπε κάποιες εκατοντάδες που για μια τόσο μικρή χώρα είναι σημαντικό και έχουμε επομένω 19 τέτοιες περιπτώσεις ε, τρομοκρατίας και, και άλλους 12 που είχαν εμπλακεί και είναι επομένω πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει στενή συνεργασία με την αστυνομία. Ε, Τη χώρα και από την άλλη μεριά όλη της αστυνομία τη Ένωσης να υπάρχει έλεγχο στα σύνορα γιατί είναι διάτρετα αυτή τη στιγμή, ιδίω όσον αφορά τα σύνορα με την Σερβία και έτσι είναι πάρα πολύ εύκολο να έχουμε εμπόριο όπλων και από του ε, φονταμεταλιστέ και από του οργανωμένου εγκληματίε. Οπότε εκεί πέρα υπάρχει όπω λένε κάποιοι αναλυτές ε, ένα διάδρομο δημοκρατίας και σε σχέση με αυτό να δούμε τι λέει και παραδείγματο 17 και εκεί τονίζεται το ότι έχουν γίνει κάποια βήματα, οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, αναφέρεται η υψηλή ανεργία της χώρας, Βέβαια, αυτά ευνοούν τους ε, ε, τρομοκράτες οι οποίοι ωφελούνται από την ανέχεια και την απληψία του πληθυσμού. Merci, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να υπογραμμίσω την υποστήριξη προς την κυρία Λούνετσεκ. Πράγματι, στο σημείο 1 αναφέρεστε ε, στο, σε άτομα που είχαν, έχουν εγκληματικό παρελθόν. Αντί αμφισβητήσιμο όπως αναφέρατε και στο σημείο 1 υπογραμμίσατε όπως έκανε και ο συνάδελφος την εγκληματικότητα στα ναρκωτικά, την τρομοκρατία και το εμπόριο ανθρωπίνων οργάνων, όπου εκεί υπήρξε και εμπλοκή των αρχών. Να υπογραμμίσω επίσης στο σημείο 5, σωστά, στο σημείο 5 λέγω σωστά, Αναγνωρίζετε ότι ανησυχείται από την έλλειψη κάθε της προόδου στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Και στο σημείο 12 επίσης αναγνωρίζεται σύμφωνα αρχή της επικουρικότητας ότι δεν υπάρχει ομόφωνη αναγνώριση του κοσυφοπεδίου. Κατά την άποψή μου, λαμβάνοντας υπόψη το σημείο σας 5 και το σημείο 1, δεν θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία ένταξης του κοσυφοπεδίου. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και την κυρία Λούνατσεκ για την περιεκτική αυτή προσέγγιση. Στο κοσυφοπέδιο υπάρχουν σημαντικά προβλήματα. Φαίνεται και είναι σαφές ότι θα πρέπει να υπάρχει εκδημοκρατισμός της χώρας οι εκλογές έγιναν με το σωστό τρόπο, αλλά άργησε ο σχηματισμός της κυβέρνησης και υπάρχει το θέμα της ίσης εκπροσώπησης των φύλων. Υπάρχουν κάποια θέματα όμως επί των οποίων θα πρέπει να μείνουμε σε ό,τι αφορά την αναγνώριση του κράτους από πέντε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά δεύτερον, μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης θα πρέπει να γίνει και ολοκληρωτική υπογραφή και σε ό,τι αφορά επίσης ε, θέματα απελευθέρωσης των θεωρήσεων θα πρέπει να εμείνουμε. Περαιτέρω, θα πρέπει να τηρηθεί το σχέδιο δράσης για τις βίζα, για τις θεωρήσεις. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να υπογράψει μια συμφωνία πλαίσιο για το να μπορεί να συμμετέχει στα ευρωπαϊκά προγράμματα προκειμένου να λαμβάνει κονδύλια από την Γεροπόλη για παράδειγμα. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό και πιστεύω ότι και η εφαρμογή των υφιστάμενων συμφωνιών είναι απαραίτητη όπως για παράδειγμα η συμφωνία μεταξύ Βελγαδίου και Πρίστινα αλλά και άλλων συμφωνιών ε, από το 2013. Επιπλέον θα ήθελα να τονίσω ένα μικρό παράδειγμα. Στο βορρά της Μητροβίτσα υπάρχει μια γέφυρα που σκοπό είχε να επιτρέψει την ελεύθερη διέλευση ατόμων και εμπορευμάτων. Νομίζω ότι θα πρέπει να βρεθεί μια λύση μεταξύ των δύο χωρών. και Σερβίας. Σε κάθε περίπτωση όμως καλωσορίζω την πολύ καλή αυτή εκθέση. Ευχαριστώ και εγώ θέλω να επενέσω την κυρία Λούνατσεκ. Πάρα πολύ καλή συγγήτρια και χαίρομαι που συνεχίζει να παίζει αυτό το ρόλο. Όπως και ο κύριος Παντζέρη πρέπει να πω ότι η ομάδα μας ε, είναι ικανοποιημένη με το κείμενο που μας έδωσε. Το νέο κοινοβούλιο σαφώς θα πρέπει να πετύχει συνένεση όσον αφορά την αναγνώριση. Ελπίζω η προτινόμενη διατύπωση να στηριχθεί από την Επιτροπή και από το Κοινοβούλιο. Θετικότατες οι προτάσεις της. Ο τηλεφωνικός κώδικας είναι πολύ σημαντικός, είναι σημαντικός ο συμβολισμός. Και αυτά που λέει για την πρόοδο όσον αφορά τον βορρά του Κωσυφοπεδίου είναι σημαντική διατύπωση που ενθαρρύνουμε τη συνέχεια της προόδου μεταξύ Σερβίας και Κωσυφοπεδίου και όλοι θα δώσουμε τροπολογίες και θα προσπαθήσουμε να βρούμε συνενετικές λύσεις. Θέλουμε να δημιουργηθεί ένα θετικό περιβάλλον για την επίτευξη πρόοδου, για την Ιούλεξ και τη διαφθορά. Εγώ ζήτησα να τεθούν σκληρά ερωτήματα και σωστό είναι να το κάνει η Επιτροπή μας. Πρέπει να σημειωθεί πρόοδος πριν ψηφιστεί στην Επιτροπή και στην Ολομέλη έκθεση. Συμφωνεί κυρία Λούνατσε και εσείς κύριε Μπροκ ως Πρόεδρος Επιτροπής. Σας στηρίζει και η ομάδα μου. Πρέπει αυτό να εξασφαλίσουμε, αυτό να συμβεί τελικά, στον αφορά τη στήριξη της έκθεσης. Εκτός μικροφώνου, κ. Μπρόκ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω και την κυρία Λούνατσα και τις προσπάθειες που κατέβαλε για την υποστήριξη της προσπάθειας για ένταξη που καταβάλει το Κωσυφοπαίδιο. Να τονίσω εκ νέου, το Κωσυφοπαίδιο είναι μία από τις στοχότερες χώρες στην Ευρώπη. Οι νέοι κυρίως μαστίζονται την ανεργία. Και δεν έχουν πολλά περιθώρια για δουλειά οι νέοι. Και έτσι μπορεί να ανθίσει το οργανωμένο έγκλημα στη χώρα. Άρα πρέπει να βοηθήσουμε τις αρχές του Κωσυφοπαιδίου να καταπολεμήσουν το φαινόμενο. Και η νέα κυβέρνηση ελπίζουμε ειλικρινά να προωθήσει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα σχετικά με αυτό. Ευπρόσδεκτες οι εκκλήσεις που ακούστηκαν για την ε, φιλελευθεροποίηση του καθεστώτος για χορήγηση θεωρήσεων για το σωποπεδίο. Θα πρέπει γρήγορα να εξασφαλίσουμε ότι οι νέοι, εκείνοι που είναι φτωχοί, χωρίς λεφτά, να μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα. Είδε μη ε, βοηθάμε το οργανωμένο έγκλημα να ε, αναπτύσσεται ανασφάλεια στα σύνορα προωθείται η παράτυπη μετανάστευση και το εμπόριο ανθρώπων. Ελπίζουμε φέτος να προχωρήσει το κοσυφοπαίδιο για να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Και εγώ συμμερίζομαι την ανησυχία της κυρίας Λούνατσεκ όσον αφορά τη χαμηλή εκπροσώπηση των γυναικών στην κυβέρνηση. Νομίζω ότι αυτή η προσέγγιση δεν αντιπροσωπεύει μια σύγχρονη κοινωνία. Ελπίζουμε να αλλάξει η κατάσταση να υπάρξει μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των φίλων. Τέλος, εκτιμώ τα μάλα την ανοιχτή έκκληση προς τα πέντε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να αναγνωρίσει το κωσυφοπεδιο ειναι Είναι σημαντικό αυτό. Χρειάζεται εξομάλυνση σχέσεων Σερβίας-Κοσυφοπεδίου. Να συνεχιστεί ο διάλογος. Ελπίζουμε στις 9 Φεβρουαρίου όταν συναντηθούν οι δύο πρωθυπουργοί στις Βρυξέλλες να επιτευχθεί πρόοδος. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Λούντσεκ, συνάδελφε, συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με όσα λέει η συγκεντρία. Νομίζω ότι το ψήφισμα πιστά αποδίδει την πρόοδο της χώρας κατά το 2014 για την Συμφωνία Σταθερότητος και Συμφωνία σύνδεση όσο γίνονται στον διάλογο για την διόρυση διαβατηρίου, τη χαλάρωση των μέτρων, όσα βγήκαν από την έρευνα της Task Force, γίνονται συνεχώς αλλαγές στη χώρα και πολύ σωστά καλυφθήκατε τη συζήτηση η κατάσταση οικονομική και κοινωνική στη χώρα. Τονίστηκαν αυτά τα οποία απασχολούν το Κοινοβούλιο αλλά και την Επιτροπή για το κράτος δικαίου, τα δικαιώματα και το να υπάρξει τελικά ε, συγκεκριμενοποίηση, να υπάρξουν απτές αποδείξεις πρόοδου για τη δικαιοσύνη και το έγκλημα. Είδαμε τι έχει γίνει από τον ε, Ιούλιο, το κείμενο των υπαντεύσεων ε, πρόκειται τους αμέσως μήνε να δημοσιοποιηθεί απλώ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζουμε ότι όλα θα προχωρήσουν γρήγορα και ότι θα επανέλθουμε εδώ και με ε, τη διαδικασία τη Συμφωνίας γνώμη θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε για τη συμφωνία με τη χώρα και μόλις τεθεί σε ισχύ η χώρα τότε δεν θα χρειαστούν τίποτα ενδιάμεση συμφωνία ή άλλου είδου διαδικασίε κυρώσεων. να ε, συνεχιστεί το ίδιο θετικό πνεύμα διαπραγμάτευση με τη χώρα. Ευχαριστώ, λέει η συγκίτρια. Άμα δεν άφησε το μικρόφωνο δεν μπορώ να ακούσω ότι μου δίνει το λόγο, αλλά τέλος πάντων ευχαριστώ όσους ε, μίλησαν, ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Συμφωνούμε, πάντως υπάρχει δημοκρατία στο Κοινοβούλιο. Και εσείς κύριε Περίρα, όταν λάβετε το λόγο, κύριε Πρέντα, κύριε Πρέντα, ως ε, συντονιστής του ΕΛΚ, ε, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ότι συμφωνήσατε. Έτσι το βλέπω κι εγώ. Ήταν πολύ θετικό ότι συμφωνήσατε, αλλά δεν συμφωνήσατε για το ότι υπάρχει πάντως ε, ε, κάποιο είδου ε, ε, κάποιο προπόθεση μεταξύ πρόοδου συμφωνία και αναγνώριση του πεδίου. Πάντω θα πρέπει και αυτό το θέμα να προωθεί μέσα από τον διάλογο ε, και να μπορέσει τελικά η Σερβία να έχει την ευκαιρία να, να δει αυτό το οποίο όλοι οι άλλοι έχουν αναγνωρίσει. Επομένω, ε, νομίζω πρέπει η διατύπωση του κειμένου να μείνει όπως την έχω εγώ και για την Ιούλεξ. Πολλοί από εσά ανέφεραν το πρόβλημα ότι δηλαδή θα πρέπει να έχει περισσότερε αρμοδιότητε, να εμπλακεί περισσότερο, να σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο. Κοίταξε την αμέσω προηγούμενη εβδομάδα. Έγινε πρόοδο. Μετά δύο χρόνια είχαμε από την εισαγγελία τις πρώτες καταγγελίες διαφθοράς σε σχέση με τον φορέα ιδιωτικοποίηση στη χώρα. Επομένω, να που η Ιούλεξ κάνει το πρόοδο. Νομίζω ότι αυτό δεν συγκροτήθηκε η Ιούλεξ. Έχει σημειώσει πρόοδο. Είναι αλήθεια βέβαια, εμεί θα θέλαμε να έχει κάνει περισσότερο και το θέλουν και πολλοί στο περίοδο. Κύριε Βότμαν, ευχαριστώ. Είστε νέα στην Επιτροπή μας. Όχι, όχι, δεν απαντώ σε όλους. Απαντώ μόνο σε όσους ρώτησαν κάτι συγκεκριμένο. Όντως, θα πρέπει να δούμε περισσότερο το θέμα των επενδύσεων, των ε, ε σχέσεων. Τώρα τον κύριο Καστάλτο. Από ό,τι γνωρίζω κύριε Καστάλτο, έχει ψηφιστεί ο νόμος για τους ξένους μαχητές. Και όσον αφορά τους ελέγχους στα σύνορα, εάν η Σερβία να γνωρίσει το Χρυσοπαίδιο θα βοηθήσει και αυτό, γιατί τώρα τα σύνορα της χώρας δεν έχουν διεθνή αναγνώριση, άρα θα βοηθηθεί και η καταπονήση της τρομοκρατίας. Όταν επικοινωνώ την κυβέρνηση, φασίζουμε στο ότι θεωρώ ότι η αφετηρία βάση είναι η αναγνώριση της χώρας. Δεν ξεκινάω το ότι υπάρχει εκεί κάποια εχθρότητα. όπω είπαν κάποιοι συνάδελφοι. Η συνάδελφος από την Κροατία, νομίζω, ή ο συνάδελφος. Από ό,τι κατάλαβα, είπατε ότι δεν υπάρχει ισότητα δύο φίλων στη χώρα. Κοιτάξτε, έχουν εκλογικό νόμο στη χώρα που προβλέπει το 30% των να είναι γυναίκες. Τουλάχιστον 30%. Εγώ επέκρινα την, την κυβέρνηση ότι δεν αποτελείται από και από γυναίκες τέλος πάντων ενώ υπάρχουν τόσες αξιόλες προσωπικότητες στη χώρα. Κύριε Υπαρκή, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα οποία είπατε για την ASA και εγώ ελπίζω να υπάρχει πρόοδο στο μέλλον. Παρακαλώ όλοι και εσείς οι σκιοδοσηγητές να αποβάλλετε τροπολογίες να καταλήξουμε σε κάποια βελτιωμένη έκθεση, όπως εσείς θα την βελτιώσετε. Και όπως είπε Μακάλιστερ, 27 πρώτου το μεσημέρι είναι η καταληκτική προθεσμία για τις τροπολογίες. Σας ευχαριστώ και τώρα περνάμε στο σημείο 9. να τονίσω ότι είχα προτείνω, ότι είχα προτείνω το έγγραφο εργασία αυτή η ετήσια έκθεση όπως ε, συζητήθηκε. Δεν θα πρέπει να καταρτίζεται στο πλαίσιο μιας έκθεσης roundabout. Για να περιλαμβάνουμε όσο έχει πολλά κράτη γίνεται, αλλά θα πρέπει να εστιαζόμαστε σε κάποια θέματα. Αυτό να το λάβετε υπόψη για τις τροπολογίες σας. Ξέρω ότι διάφοροι πρεσβευτές θέλουν να στραφούν στους συναδέλφους προκειμένου να μπορούν να το παρουσιάσουν μετά στην πατρίδα τους ως επιτυχία ότι να συμπεριληφθεί σε και αυτή η πρόταση. Δεν είναι αυτός ο στόχος της έκθεσης. Να ληφθεί σας παρακαλώ υπόψη ότι εδώ προσπαθούμε να θέσουμε κάποια γενικά μηνύματα να αποστείλουμε ως απάντηση στην ετήσια έκθεση της ΥΠΑ της εκπροσώπου και αντιπροέδρου. Έγινε μια συζήτηση με τα εθνικά κοινοβούλια και κάποια εθνικά κοινοβούλια κατέθεσαν προτάσεις τις οποίες εν μέρη λάβαμε υπόψη. Θα ήθελα και θα ήμουν ευγνώμων να υποβάλλετε τις προτάσεις σας το συντομότερο δυνατόν για να τις λάβουμε υπόψη. Επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ καιρό, είμαι δεσμένος να το συζητήσουμε και στις 26-27 ή το θέμα αυτό περαιτέρω. Δεν το συζητήσα με τη γραμματεία ακόμα, αλλά ελπίζω να μην μου θυμώσει η γραμματεία. προκειμένου και μετά τη συζήτηση να έχουν τη δυνατότητα οι συνάδελφοι να κρατήσουν τροπολογίε. Η έκθεση τώρα ξεκινάει με μια σύντομη παρουσίαση τη κατάσταση σε ό,τι αφορά τη γεωπολιτική ασφάλεια, την οποία έχουμε σήμερα σε παγκόσμιο στο προσκήνιο αυτό. Και εκεί λοιπόν προσπάθησα να επικεντρωθώ σε τρει προτεραιότητε. Καταρχά, για την ενίσχυση των ικανοτήτων μας να μπορούμε να αντιδρούμε στην παγκόσμια σκηνή αποτελεσματικά βελτιώνοντας τις εταιρικέ διεργασίες και τις διαθεσμικές μας ε, διεργασίες. Και προς την κατεύθυνση αυτή θεωρώ ότι δεν έχουμε ακόμα πλήρως αξιοποίηση τη συνθήκη της Λισαβόνας, ε, κοιτώντας τι γίνεται με τις πολιτικές για την εξωτερική και την εσωτερική πολιτική και οι δύο έχουν μια ισχυρή εξωτερική διάσταση και θα πρέπει από κοινού να θεωρούνται. Και μιλώντας για θέματα χρηματοδότησης θα πρέπει να κοιτάξουμε τα δημοσιονομικά μας μέσα γιατί αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα. Θεωρώ ότι όλο το σύστημα θα πρέπει να διαμορφωθεί με πιο ευαρύτη τρόπο και με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Επίσης, θέματα και της συνεργασίας, το θέμα της άμυνας, εν ώψη και της μελλοντικής συνόδου. Θα υπάρξει μια ξεχωριστή όμως έκθεση για τα θέματα αυτά σε ό,τι αφορά την ε, πολιτική ασφάλειας. Δεύτερο στοιχείο. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να παρουσιάσουμε το ότι η ευρωπαϊκή πολιτική, ε, πολιτική τάξη θα πρέπει να διασφαλίζει την νομική τάξη. Αυτό συζητιέται σε σχέση και με την ε, γειτονία προς Ανατολά, θέματα αναλογικότητας, επικουρικότητας, ε, θεμελιωδών ανθρωπινών δικαιωμάτων. Αυτά θα πρέπει και με πολιτικό και οικονομικό τρόπο να υποβοηθούνται. Τρίτος τομέας οι εξελίξει στην γειτονιά προ τον Νότο. Σταθερότητα και ασφάλεια. Ξέρουμε ότι τα πολιτικά και οικονομικά συστήματα θα πρέπει να εξυγχρονιστούν και εμεί όμω θα πρέπει να συμβάλλουμε προκειμένου να τερματιστούν οι ενόπλες σειράξεις και σε συνεργασία με τους διεθνεί, αλλά και με τους περιφερειακούς φορείς. Το τελευταίο θέμα έχει να κάνει με την ε, διεθνή δημόσια τάξη και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη εργασία μας με τη ΣΥΠΑ και με το ΝΑΤΟ. Αλλά υπάρχουν και σημαντικά θέματα τα οποία θα πρέπει να τα κοιτάξουμε με την Κίνα, για παράδειγμα, με τη Ρωσία, όπου θα πρέπει να διασφαλίσουμε την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά από την άλλη είμαστε έτοιμοι να αναζητήσουμε οδούς επικοινωνίας προκειμένου από κοινού να φέρουμε την ευθύνη για την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα. Ελπίζω αυτή η προσέγγιση να σας βρει σύμφωνο και θα χαιρόμουν με μια συζήτηση επί του προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η έκθεση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Η κυρία Λούζικ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όπως για πολλές εκθέσεις και για την έκθεση αυτή θα πρέπει να πω ότι σε κάποια ζητήματα είμαι λίγο διστακτική. Πολλά ζητήματα από δικής μας πλευράς πρέπει να πω ότι τα αξιολογούμε θετικό τρόπο, όπως για παράδειγμα η προσέγγιση ότι ο εισηγητής ε, θέλει μεταρρύθμιση της μεταναστευτικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα εστιάζεται στα πραγματικά αίτια της μετανάστευσης τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ότι ζητάει τον τερματισμό κρίσεων και πολέμων και καλή όλους τους φορείς όπως το, τη Ρωσία, την Κίνα, το Ιράκ και άλλους περιφερειακούς φορείς να συνεργαστούν. Πολλά είναι θετικά λοιπόν. Σε ό,τι αφορά την επιδείνωση του πλαισίου ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρούμε ότι αυτό πάντα αποτελεί ζήτημα ε, αιτιαού και αιτιατού. Στην έκθεση αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε καμία περίπτωση δεν έχει εξαντλήσει τις δυνατότητες ε, που έχει στα χέρια της. Θεωρώ ότι έχει εξαντλήσει παρόλα αυτά πολλές δυνατότητες η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ερώτημα είναι τι αποτέλεσμα, τι αντίκτυπος υπάρχει. Και το αποτέλεσμα είναι ότι τελικά τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από ό,τι στην αρχή σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της πολιτικής, του δυναμικού. Κοιτώντας για παράδειγμα την γειτονία με τις χώρες του Νότου. Η επιρροή στις οικονομίες των χωρών της ε, γειτονίας προς τον Νότο ήταν αρνητική. Αποσταθεροποίηση. Οικονομική. Αυτό αφορά και πολιτικά ζητήματα, αλλά και θέματα ασφάλειας. Δεν νομίζω ότι είναι ποσοτικό μόνο το ζήτημα. Δεν χρειάζεται μόνο δηλαδή ποσοτική εξάντληση των μέσων. Μιλάμε και την, για τη θεμελιώδη πολιτική κατεύθυνση, τον πολιτικό προσανατολισμό των μέσων. Εδώ θεωρώ ότι υπάρχει μια διαφωνία επί της αρχής. Όπως και σε θέματα εμπορικής πολιτικής, πολιτικής εξωτερικών υποθέσεων, πολιτικής ασφάλειας. Εδώ είναι αφήσει οι διαφορές που έχουμε στις ε, τοποθετήσει μας. Άλλο ένα ζήτημα θα ήθελα να θίξω συγκεκριμένα. για την απλοποίηση της διάθεσης κονδυλίων σε ό,τι αφορά τους ε, αντιπροσώπους, ε, τους επικεφαλής των αντιπροσωπιών. Ένα, ένα θέμα θα αναφέρω μόνο, Πρόεδρε. Αυτό αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι αφορά τον έλεγχο προπολογισμού στα πλαίσια της δημοσιονομικής πολιτικής και του δημοσιονομικού δικαίου, όπου δίδονται καλές ε, δυνατότητες ε, στο Κοινοβούλιο Στο Κοινοβούλιο τα συζητήσαμε αυτά και την προηγούμενη εβδομάδα. Και θα ήθελα πιο πολύ πίεση να ασκηθεί στην Τουρκία. Αυτό στην έκθεση δεν αναφέρεται παρκώς. Θεωρώ ότι είναι έκθεση μειονότητας λοιπόν συνοπτικά αυτή η έκθεση. Σα ευχαριστώ πολύ. Αλλά το θέμα αυτό δεν έχει τεθεί εξίσου στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Κούκαν. Ευχαριστώ δύο συντόματες παρατηρήσεις. Η έκθεση ίσως έχει είναι καλή. Και μετά από την έκκλησή σας για τροποποίησή της, νομίζω ότι άμα γίνουν αυτές οι αλλαγές θα έχουμε σημαντικότατο έγγραφο. Θέλω να εκφράσω πλήρη υποστήριξη όσον αφορά την φιλοσοφία της εκθέσεως που μας εξηγήσατε, αυτό που προτείνατε, να μπούμε σε λεπτομέρειες όσον αφορά τις χώρες θέλουμε μια γενική προσέγγιση για το έγγραφο που θα περιέχει συμπεράσματα και θα εξυπηρετεί το σκοπό καθορισμού καθατευθυντήριων γραμμών για την εξωτερική μας πολιτική, για την αντιμετώπιση του σημαντικότατου ζητήματο. Θα πρέπει αυτά τα χαρακτηριστικά να διατηρηθούν όσον αφορά το κείμενο. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ο κ. Μποστινάρου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαιρετίζω τη συνεισφορά σας και επαναλαμβάνω ότι στη στατηγική να αναφέρουμε ότι χρειάζεται σχετισμός και συντονισμός μεταξύ ασφαλείας εξωτερικής πολιτικής και άμυνας μαζί με την ενεργειακή πολιτική. Η για τη μελλοντική ε, ενεργειακή ένωση πρέπει να ε, κινηθούμε. Ο κ. Σεύσοβιτς προχθές συνάντησε τον Αλεξέη Μίλα από την Gazprom και έθεσε το νέο κίνδυνο, δηλαδή η Ρωσία να περιορίσει τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης. Θα πρέπει να αναφερόμαστε ρητά στην ανάγκη συσχετισμού και συντονισμού μεταξύ των πολιτικών, διότι σήμερα ενέργεια ίσον ε, ασφάλεια για την Ένωσή μας. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το σχέδιο ψηφίσματος. Ε, περιέχει διάφορες παρατηρήσεις, σωστές παρατηρήσεις, κυρίως το, το σημαντικότερο για τη συνεργασία μας στην εξωτερική πολιτική είναι να θεσπίσουμε ένα στρατηγικό στόχο, στόχους που θα πρέπει να επιδιώκουμε από κοινού. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε και το εξής. Δηλαδή, ανάμεσα στους στόχους αναφερόμαστε στην ασφάλεια των ευρωπαϊκών χωρών, των κρατών μέλων, επίσης του Νότου. Αναφερόμαστε στη Νότια Ευρώπη. Όμως, θα ήταν ίσως καλύτερο να πούμε ότι κοινό στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έπρεπε να είναι η στήριξη της ανεξαρτησίας των χωρών που απέρευσαν από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Κοιτάξτε, τι... αυτό βέβαια συνέβη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πολλές από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης αποτελούσαν κομμάτι της Σοβιετικής Ένωσης παλιά. Και οι μισές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν δεδομένη την ανεξαρτησία τους για πάντα. Αυτό θα πρέπει να το αναφέρουμε όσον αφορά τη συνεργασία. Κάποια χρόνια πριν, όταν αναφερόμενοι στη χώρα μου μιλήσαμε για ένα σύνταγμα για την Ευρώπη, τότε που συζητούσαμε τη συνθήκη της Λισαβόνας, ένας από τους στόχους για την εξωτερική πολιτική τότε θα ήταν να τίθενται κοινή στόχοι. Πρέπει να προσέξουμε το αρχικό κομμάτι που λέμε ότι θέλουμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας και τις αρμοδιότητες καθορίζοντας κοινού στόχους. Θα πρέπει να δούμε και προς Ανατολά στον αφορά τους στόχους. Χρειάζεται διεθνή συνεργασία. Και στα πλαίσια της συνεργασίας χρειάζονται θεσμοί για την επίτευξη των κοινών συμφερόντων και των κοινών στόχων. Πρέπει να αναπτύξουμε τους αναγκαίους θεσμούς. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Αγαπητοί συνάδελφοι, ναι, πρόκειται σαφώς για ποιοτική έκθεση. Και μάλλον είναι επικέστριο το το στην να την έκθεση εφαρμογής για την ε, την έκθεση για την εφαρμογή της, της πολιτικής ασφάλειας στην ΣΕΝΤΕ στην Υποεπιτροπή για την Ασφάλεια. Γιατί εδώ πέρα τώρα έχουμε το θέμα της τρομοκρατίας. Η τρομοκρατία δεν αναφέρεται πουθενά. Και επίσης ε, στην έκθεση Συμβουλίου και Επιτροπής, ακροφυγός μόνο αναφέρεται. Όμως βλέπουμε ότι τη σημερινή μέρα είναι κάτι το πάρα πολύ επίκαιρο. Και πρόκειται για ένα κίνδυνο θα πρέπει να τονιστεί αυτός ο κίνδυνος και επίσης θα πρέπει να τονίσουμε τη δυνατότητα Ένωση και κρατών μελών να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία. Άρα, να τονιστείτε ότι χρειάζεται καλύτερο συντονισμό και καλύτερη συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη για όλα αυτά, για ασφάλεια δηλαδή και εξωτερική πολιτική. Μέχρι τώρα δεν έχουμε αρκετή τέτοια συνεργασία. δεν έχουμε αρκετές πληροφορίες όσον αφορά τα θέματα ασφάλειας. Τώρα, κάτι άλλο. Συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Είναι κάτι που είναι αρμοδιότητά τους μέχρι σήμερα. Ε, γι' αυτό και χρειάζεται συνεργασία. Μέχρι τώρα είχαμε σαν πλατφόρμα συνεργασίας τη διάσκεψη για ασφάλεια και εξωτερική πολιτική που ε, την, γνωρίζουμε ως Κόζακ. Και πρόκειται για έναν παράγοντα που αναφέρεται και αυτό στην έκθεση. Thank you, Chair. Uh, we would also like to stress that we consider... Πρόεδρε, να τονίσω ότι είναι πολύ ισορροπημένα τόσο άλλη έκθεση. Δεν επισερχόμαστε στις λεπτομέρειες. Λέμε τα πιο κρίσιμα ζητήματα, ασφάλεια συνόρων, εξωτερική πολιτική. Να, δύο σημεία που θέλω να σας αναφέρω. Πρώτα πρώτα, ότι θα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο τις προοπτικές που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, δεν λέει και πάρα πολλά η έκθεση, αλλά δεν πειράζει. Όμως, όμως θα πρέπει να επισύρω την προσοχή σας σε κάτι το οποίο αποτελεί μια πρόταση. Στο πώς τα ανθρώπινα δικαιώματα θα ενταχθούν σε κάθε ζήτημα εξωτερικής πολιτικής όχι μόνο στην ενεργική πολιτική, αλλά και στην εμπορική πολιτική και στην αναπτυξιακή πολιτική. Θα σας υποβάλουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Σα uh, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θεωρώ ότι η να αναγνωρίζει επαρκώς το γεγονός ότι υπάρχει διαφορετική προσέγγιση και πολιτική από διάφορες χώρες. Αυτή η προσέγγιση ότι μία λύση ταιριάζει σε όλους ε, είναι ένα εμπεριαλιστικό νομίζω, μια εμπεριαλιστική ένδειξη και αυτό σε ό,τι αφορά την πολιτική για την Ρωσία, για την Αργεντινή και προφανώς αυτά που έχουν συμβεί στην ε, Ανατολική Ευρώπη έχουν προκαλέσει την Ρωσία. Πώς μπορεί να υπάρχει συσχετισμός για τέτοια θέματα όταν βλέπουμε ισπανικές εχθρότητες και ε, τις δράσεις που συνεχίζονται στο Κεβραλτάρι, για παράδειγμα. Ευχαριστώ. Then we have Mr. Merci beaucoup. Κύριε Πρέντερ, ευχαριστώ κύριε Πρέντε. Mm. Καταρχάς να σας συγχαρώ για την ε, έκθεση αυτή που έχει μια γενική προσέγγιση που υποστηρίζει το ΕΛΚ. Θα ήθελα και εγώ να πω ότι συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Κούκαν για τις τροπολογίες και με αυτά που είπατε στην αρχή ότι θα πρέπει να κρατήσουμε το μορφότυπο αυτό και να μην επισέλθουμε σε υπερβολικές λεπτομέρειες. Θα ήθελα επίσης να εμείνω στο γεγονός ότι μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε τον τόνο που προτείνεται και από αφενός για να θέσουμε τα θέματα των συμφωνιών με τη Μολδαβία και την Ουκρανία σε ό,τι αφορά και την προετοιμασία μελλοντική προσέγγιση με την Ένωση και από την άλλη το γεγονός ότι ε, αναφέρεται τις σχέσεις με τη ΣΥΠΑ. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και θα πρέπει να παραμείνουμε στην φιλοσοφία αυτή την οποία προτείνεται. Οι συνάδελφοι που έχουν ε, ως σήμα κατά τεθέν τον αντιμερικανισμό θα ήταν κρίμα να ικανοποιηθούν σε αυτή τη φάση γιατί θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες με τη ΣΥΠΑ και θα πρέπει να ολοκληρώσουμε και τις διαπραγματεύσεις για το Ευχαριστώ. Well, uh, the report is uh, solid. Η έκθεση είναι σίγουρα πολύ καλή και πολύ καλογραμμένη. Και επειδή είναι γενικά η γενική συζήτηση, θα πρέπει να έχουμε κατά νου το έργο τη είπα τη εκπροσώπου νομίζω ότι μπορεί να διαρρεθεί σε δύο τμήματα. Καταρχά, να φροντίσει όλα τα θεσμικά όργανα και όλα, όλες τις υπηρεσίες που υπάγονται στον τομέα των αρμοδιοτήτων της και θα πρέπει να βελτιώσει τη λειτουργία τους, αλλά αφετέρου και ίσως και πιο σημαντικό πρέπει να αποτελεί και ενδιάμεσο διευκολυντή της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών. Και εδώ νομίζω ότι είπα ότι εκπρόσωπος πραγματικά μπορεί να διαδραματίσει το ρόλο που θα συγκεντρώσει όλες τις ε, τοποθετήσεις, στα... ξεκινήσει πρωτοβουλίε όπω και προβλέπει η συνθήκη τη Λισαβόνα. Και εδώ θεωρώ ότι θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί ιδιαίτερα και αυτό θα πρέπει να αποτυπώνεται και στην έκθεση. Αποτυπώνεται μεν, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να δοθεί περαιτέρω έμφαση στη διάσταση αυτή ακριβώ. Και εγώ, Πρόεδρε, να συγχαρώ. Ποια δουλειά που έκανε. Φιλόδοξο κείμενο και πολύ πλήρες. Πρόκειται για περίπλοκα σημεία. Το διεθνές περιβάλλον διεθνή συγκυρία είναι περίπλοκη. Τονίζει το ρόλο της υπάρξης εκπροσώπου. Το ζήτησε αυτό το Συμβούλιο και νομίζω ότι όσα είπες είναι χρήσιμα στην υπατή εκπρόσωπο. Χρειάζεται συντονισμός, χρειάζεται συνεπίσταση ένωση και κρατών μελών για την πολιτική άμυνας και ασφαλείας. Πολύ κρίσιμο τόσο ελέγχθησαν επίσης για τις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάτι να πούμε για την ε, Λιβύη. Εγώ θα καταβάσω μια τροπολογία. Ο ΙΕ καταβάλει προσπάθειες. Έγιναν και επαφές στην Γενέβη, όπως γνωρίζουμε πρόσφατα. Να δούμε τι θα γίνει με τη συνάντηση του Ιουνίου. Παράγραφος 35 αφορά την βία του χαλιφάτου, της τζιχάντ. Θα πρέπει επίσης να δούμε τι γίνεται με την παράγραφο 40 και την 41. Είναι και το, εκεί το θέμα του κλίματος, αλλά τέλος πάντων θα πρέπει να αναφερθούμε περισσότερο στην διεθνή τρομοκρατία. Και Πέραν του, της του κλίματος και της, και της ε, συνθήκης μη διάδοσης των πυρηνικών, λέει ξανά, Σπέραφο 35 ίσως, ή κάπου, τέλο πάντων, να εντάξουμε μία προσθήκη για την τζιχάντ. <clears throat> Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόσφατα εστιαστήκαμε επί της ανάγκης κοινή ενεργειακής πολιτικής. Σαφές μήνυμα για όλους μας. Πρέπει και στην πράξη να εφαρμόσουμε αυτές τις αποφάσεις. Πετύχαμε πολλά. Σωστά αναφέρθηκε ότι χρειάζεται προβληματισμός επί των επιτεγμάτων και μελλοντικών προκλήσεων. Ας εισερθούμε τώρα, Πρόεδρε, στην παραπληροφόρηση και την προπαγάνδα και τη σχετική πολιτική. Την Πέμπτη, την περασμένη εβδομάδα, εγκρίναμε ψήφισμα για την κατάσταση στην Ουκρανία. Και στο κείμενο γινόταν έκκληση προς τον Επίτροπο Χάν να ετοιμάσει κάποιο έγγραφο σε δύο μήνες. Αυτό είναι πολύ επίκαιρο. Και στο ψήφισμά μας πρέπει να αναφερθούμε στην ανάγκη για γενικότερη αποτελεσματικότερη πολιτική ενημέρωσης. και αυτά στα πλαίσια της πολιτικής ασφαλείας. Θα κάνουμε σχετικές προτάσεις για το έγγραφό σας που είναι άριστο και ελπίζουμε να συμφωνήσουμε. Να συμφωνήσουμε επιτυχών προσθήκων στο κείμενο για τις επόμενες ημέρες. Συνεχίζει χωρίς μικρόφωνο ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Με τη σειρά μου να σας συγχαρώ για την κατεύθυνση της εκθέσεως. Πέρα από τις τροπολογίες που θα καταθέσω, αν μπορούμε να επιμείνουμε επί τεσσάρων σημείων. Πρώτον, καταπολέμηση τρομοκρατίας. Η απειλή δεν βαρύνει μόνο τη Μέση Ανατολή και το Μαγκρέμπ, αλλά αντιμετωπίζεται και στην Ευρώπη εν πρώτης. Και θα πρέπει να το πούμε σαφώς. Και κυρίως ε, την Αφρικανική Ήπειρο. Και κάτι άλλο που αναφέρεται και είναι σημαντικό. Ο ρόλος της άμυνας, της ευρωπαϊκής άμυνας όσον αφορά την καταπολέμηση του εμπορίου όπλων, ναρκωτικών και ανθρώπων. Που όλα αυτά συμβάλλουν στην ενίσχυση του τρομοκρατίου. Θα ήταν σημαντικό να υπογραμμίσουμε καλύτερα τη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Αμήνης και ΝΑΤΟ. Η Ευρωπαϊκή Άμυνα είναι ένας από τους πυλώνες του ΝΑΤΟ. Δεν πρέπει να το λησμονούμε. Είναι σημαντικό στοιχείο. Μπορεί να μας πατεύσει το ΝΑΤΟ, όμως υπέχουμε υποχρέωση να προστατεύσουμε και άλλες χώρες ε, εκτός να το δεχτούν επίθεση. Κι άλλο στοιχείο. Κάτι απαραίτητο. Να υπογραμμίσουμε, όπως έκανε και είπατε εκπρόσωπος, ότι χρειάζεται να ενισχύσουμε τα αμυντικά μέσα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Και όχι απλώς να εξασφαλίσουμε το συντονισμό αυτών. Τος μικροφόνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και από δική μου πλευρά να πω ότι και εγώ συμφωνώ με το σχέδιο τη έκθεση. Επί του περιεχομένου δεν έχω να κάνω οποιαδήποτε παρατήρηση, αλλά θα ήθελα να τονίσουμε ότι θα πρέπει να αλλάξει ίσω η δομή από το γενικό να περάσουμε στο ειδικό. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα το κεφάλαιο για την ενίσχυση της συνεργασίας ε, σε παγκόσμιο επίπεδο σε σημεία 37 41 να μπουν στο 22, πριν το 22, γιατί είναι η γενικότερη προσέγγιση και να υπάρχει μια αναδιάθρωση στα δύο σημεία που έχουν να κάνουν με την πολιτική προς ε, τον Νότο και να μπουν σε άλλους τίτλους, γιατί στους άλλους τίτλους, στα γερμανικά τουλάχιστον, όπου μιλάμε για τη διαφύλαξη του νομικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι θεωρώ κάπως παραλαπανητικό, γιατί μετά αναφέρεται η πολιτική προς Ανατολάς και για την προς Θεωρώ ότι λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει ένα κεφάλαιο για την ενίσχυση της πολιτικής των χωρών ε, προς τον Νότο, 32-36, αλλά ήθελα να γίνει ένα κεφάλαιο για τις νέες ε, προσεγγίσεις από το 25 έως 28 σε ό,τι αφορά δηλαδή την Ανατολή. υπάρχει δηλαδή μια ταξινόμηση αναπολιτική για τον Νότο και για την ε, Ανατολή και για τον Νότο. Να υπάρχουν ίσα-ίσα τα σημεία 28 μέχρι 32 που αφορούν τη Ρωσία να αναφερθούν ξεχωριστά για τη Ρωσία και μετά να υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο το θέμα της ε, προσχώρησης, το σημείο 23 δηλαδή. Εδώ θεωρώ μπορεί να συμπεριληφθεί αυτό το ένα και μόνο σημείο για να είναι πιο σωστέ ότι κινούμαστε από το γενικό στο ειδικό. Αυτές είναι οι διαφορετικές ε, τροπολογίε που έχω να κάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γκάλο που με βοηθάτε να καταρτήσω την έκθεση, αλλά να σας πω και ποια λογική θεωρώ εγώ ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή στην έκθεση, εν πάση περιπτώσει. Κυρία Γκάμπριελ, έχετε το λόγο στην τελευταία. Ευχαριστώ και εγώ πρόεδρε να ευχαριστήσω και να συγχαρώ Σωστά τα λέτε και με ακρίβεια. Θέλω να σταθώ σε τέσσερα σημεία. Πρώτα-πρώτα κάτι θεσμικού, λειτουργικού χαρακτήρα, για το οποίο ήδη το έναφετε στην έκθεση. Πρώτα-πρώτα του ειδικού εκπροσώπου. Χρειάζεται να του εντάξουμε περισσότερο στην υπηρεσία εξωτερική δράση. Και επίση χρειάζεται να προβληθεί περισσότερο το έργο του. Είναι περισσότερο από αναγκαίο αυτοί οι διάφοροι ειδικοί εκπρόσωποι, περιφερειακοί κλπ. να ε, προβάλλονται και να είναι σημείο αναφοράς. Και επίσης συμφωνώ με αυτό το οποίο είπατε για να διευρυνθεί η χρήση της ε, επιταχυμένης ταχείας διαδικασίας για την απεμπλοκή πόρων. Αυτό χρειάζεται για τις κρίσεις. Έχουμε πολλές ανθρωπιστικές κρίσεις ολόγυρα που είναι αποτέλεσμα πολιτικών κρίσεων. Πρώτα-πρώτα όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι να φύξουμε περισσότερο στην έκθεση για τα πολέμηση του ριζοσπαστικοποίησης της θρησκευτική και της τρομοκρατίας. Θα πρέπει οι εταιρικέ μας σχέσεις με τις βεντσουκτών προσμόντων να ενισχυθούν. Το είδαμε αυτό. Να έχουμε εταιρική σχέση η οποία να εξελιχθεί. Στενή συνεργασία με περιφερειακές ε, ε περιφερειακούς φορείς, αραβικό σύνδεσμο κλπ. Αλλά και προς Ανατολάς να γίνει το ίδιο. Και έτσι να μπορέσουμε να καταπονήσουμε την τρομοκρατία. Να συγκρατηθεί αυτό το φαινόμενο τώρα για την θρησκευτική ριζοσπαστικοποίηση, να ασχολούμε περισσότερο με αυτά τα οποία κάνουν οι εταίροι μας όπως το Μαρόκο. Πρόκειται για κάποιες πρακτικές που θα μπορούσαμε και εμείς να μιμηθούμε να υπάρχει επίση συνέπεια μεταξύ ιστορική και εξωτερική πολιτική. Στα πλαίσια αυτά υπάρχει κάτι που πρέπει να το αναφέρουμε στην έκθεση. Είναι το πώ θα υπάρχει μια αυθεντική διπλωματία μετανάστευση. Ασχοληθούμε και με τι τέτοιε χώρε του Ευρωπαίου και με μια τέτοια εξωτερική πολιτική θα μπορέσουμε να ασχοληθούμε με τις πραγματικές αιτίε του φαινομένου της παρανομής μετανάστευσης. Αλλά μπορούσαμε να καλύψουμε και την νόμιμη μετανάστευση. Άρα ας δείξουμε θάρρος να πούμε για μια πραγματική πολιτική μετανάστευση σε συνεργασία με τις τρίτες χώρες. Τις χώρες διέλευσης, τις χώρες προέλευσης. Πρόκειται για κάποιες προκλήσεις που είναι σήμερα παγκόσμιες. Um, Σα ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομο, λέει ο κύριο Χάουιτ, σε ό,τι αφορά και τα συνάδελφο ε, Πέσκο. Ε, είναι πάρα πολύ δυνατό το κείμενο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που το προετοιμάσατε. Πολλά μας βρίσκουν σύμφωνο σημαντικό ε, ρόλο τη της συνεργασία, πιο πολύ ενεργή αντιμετώπιση η ανατολική γειτονία, η θετική ανταπόκριση στην Μολδαβία, στη Γεωργία, στην Ουκρανία. Και θετικός διάλογος με τη Ρωσία. Νομίζω ότι υπάρχει και ένα τμήμα για τις κυρώσεις σε ό,τι αφορά την έμφαση στους περιφερειακούς φορείς, σε ό,τι αφορά ε, τη γειτονία προς ε, τον Νότο είναι πολύ καλαγραμμένη. Για την παράγραφο 11 θα πρέπει να το σκεφτούμε σε ό,τι αφορά την ΕΕΔ. Θα πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν πολύ ε, σωστά πώς θα πρέπει να έχει διατύπωση. Θα πρέπει επίσης να σας πω ότι συμφωνώ με την παράγραφο 12, αλλά θεωρώ ότι είναι μάλλον απαραίτητη η αναδιατύπωση, μάλλον η μεταρρύθμιση και συμφωνώ με την διατύπωση στην 12 σε ό,τι αφορά το 6 στην συνδυασμό των πόρων. Θεωρώ ότι αυτό μπορεί να παρεμεινευτεί, το ακούσαμε και από κάποιου άλλου. θα πρέπει να το κοιτάσουμε αυτό. Δεν είμαι αρνητικό στο σκοπό τον οποίο προσπαθεί να πετύχει η παραγράφο. Νομίζω ότι η κυρία Παπακερίνη είναι πάρα πολύ, ήταν πολύ σαφή για την ε, κοινοβουλευτική διαδικασία για τη μεταρρύθμιση για την εξέταση του ΚΕΠΑ στην παράγραφο 16, στην 18 για την λατρομετανάσταση. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει η πρόβλεψη για την άμεση μετανάστευση στην 20 και 21. Θεωρώ ότι η ενεργική πολιτική είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεδομένη και του Παρισιού φέτο Για την 23 δεν θα πρέπει να Δυτικά Βαλκάνια, Δυτικά Βαλκάνια και Τουρκία θα πρέπει να έλεγε. Στην 37 δεν νομίζω ότι οι διδευτικές σχέσει θα πρέπει να ορίζονται μόνο από το TTIP. όπως έχει διατύπωση και θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει μία ξεχωριστή παράγραφο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και είμαι βέβαιος ότι η ομάδα μας θα εξετάσει αυτό το ενδεχόμενο. Αλλά συνολικά είναι πολύ επικοδομητικό το κείμενο και είμαι βέβαιος ότι θα ήταν και πολύ επικοδομητική και θετική και δρασή μας σε αυτό. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι. Όντω το θέμα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας στις τελευταίες ημέρες ε, έχει ειδικό βάρος μετά τα τελευταία περιστατικά και το θέμα της σχετικής πολιτικής θα πρέπει να αναφερθούν και αν θέλετε να τα θέσουμε πιο έντονα αυτό, αν υπομονώ να ακούσω για τις δικές σας προτάσεις. Το θέμα με την, της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Σας είπα ότι και η Υποεπιτροπή θέλει να προετοιμάσει μια σχετική έκθεση, γι' αυτό δεν θέλω να τα προκαταλάβω όλα αυτά, αλλά αν έχετε κάποια πρόταση είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να βρούμε μια ισορροπημένη λύση. για να παρουσιάσουμε τις ε, απαραίτητες ε, ψυχές, όπως για παράδειγμα όταν αναφέρατε τι ανθρωπιστικέ λύσει, όταν πρόκειται για παράνομο εμπόριο όπλων, τη καταπολέμηση, τη τρομοκρατία, όλα αυτά έχουν το ρόλο του να παίξουν και εκεί. Γι' αυτό λοιπόν σίγουρα θα μα απασχολήσουν. Ευγνώμων θα ήμουν αν το συντομότερο δυνατόν μου δίνετε τι τροπολογίε σα, όχι τελευταία στιγμή αν θέλετε, για να μπορώ να κάνω και συμβαστικέ προτάσει. Να μπορούμε να κάνουμε σωστά συζήτηση και να βρούμε μια όσο πιο ισορροπημένη λύση γίνεται. Σα ευχαριστώ πολύ. Και νομίζω δεν χρειάζεται να γίνει ειδική συζήτηση στις 26 του μηνός. Περιμένουμε τις τροπολογίες σας και μετά θα κάνουμε τη συζήτηση. Και τώρα θα ήθελα να παρακαλέσω να σας αναφέρω ότι είναι, έχει ήδη καταφτάσει ο Υπουργός, αλλά είναι κυκλισμένο των θυρών η συνεδρίαση. Το δεύτερο τμήμα μόνο, διορθώνει ο πρόεδρο, είναι κυκλισμένο το θηρόν. Μόνο το δεύτερο τμήμα. Άρα ο εκπρόσωπο τη Ρωσική Πρεσβεία θα πρέπει να φύγει στο δεύτερο ημίση, λέει ο Πρόεδρο. Όχι, όχι, δεν κάνω πλάκα. Ε, είχαμε μια συνάντηση, ξέρετε, και κλεισμένο θηρεών με την κυρία Μαγκερίνη πριν τα Χριστούγεννα. Και το προσωπικό του, <laughs> της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης ήταν και ένα μέλος της ε, ρωσικής ε, πρεσβείας. Δεν σας κάνω πλάκα. That that's a sense of humor. I liked it. <laughs> Not so much. <laughs> Liebe Freunde, Αγαπητοί φίλοι, έχουμε την έκθεση του Υπουργού Εξωτερικού της Προεδρίας ε, του Συμβουλίου για την ε, πολιτική γειτονία και σε ό,τι αφορά την ε, έκθεση τη κυρία Μογκερίνη. Το δεύτερο τμήμα θα είναι κυκλισμένο το θυρών. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Sandra is your fan, I see. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ σήμερα στην συνεδρία τη Επιτροπής σα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προσβλέπω σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή και με το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια τη Προεδρία μα. Εκτιμούμε ιδιαίτερο το ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου που διαμορφώνει την εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ σήμερα για να συζητήσουμε τι προτεραιότητε τη Λετωνικής Προεδρία. Θέλω να αναφερθώ την Ευρώπη τη συμμετοχική. Είναι μια από τι προτεραιότητε προεδρία μα, μαζί με την ανταγωνιστικότητα και την ψηφιακή Ευρώπη. Και πώ θα συνεργαστούμε στενά με την Υπηρεσία Εξωτερική Δράσεω και την ύπατη εκπρόσωπο Φεντερίκα Μογκερίνη όσον αφορά τι παγκόσμιε φιλοδοξίε που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα αναφερθώ συγκεκριμένα στη διεύρυνση, ένα θέμα στο επίκεντρο τη εξωτερική πολιτική Ευρωπαϊκή Ενώσεω και κάτι που υποστηρίζω ένθερμα. Η χώρα μου πριν από 10 χρόνια εισήλθε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια δεκαετία μετά, κανεί δεν αφισβητεί τα ωφέλη τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και του καρπού των προσπαθειών. Η Λετωνία υπερασπίζεται ανοιχτή ευρωπαϊκή διεύρυνση και ανοιχτή πολιτική γειτονία. Πριν συζητήσω τη διεύρυνση, θα ξεκινήσω με κάτι που είναι λιγότερο θετικό. Που πλήττει τον ανοιχτή προσέγγιση Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σημερινή συνεδρίαση λαμβάνει χώρα όταν το διεθνές υπόβαθρο είναι πολύ σκοτεινό. Οι επιθέσεις στο Παρίσι ήταν ε, βάρβαρες πράξεις βίας και έπληξαν όλους κάθε θρησκείας. Ομή βία, δολοφονία αθώων, επίθεση κατά της ελεύθερης έκφρασης. Τα γεγονότα στο Παρίσι και στη Γαλλία έστειλαν ε, το κύμα, το οστικό κύμα σε όλη την Ευρώπη αλλά οι επιθέσεις μας ένωσαν όσον αφορά τις αξίες μας, την στήριξη της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν μας χώρισαν οι επιθέσεις, μας έδεσαν περισσότερο. Οι πορείες στο Παρίσι και σε όλη την Ευρώπη, των οποίων ηγήθηκαν οι ηγέτες, έδειξαν ότι είμαστε ενωμένοι. Ότι είμαστε αποφασισμένοι να πολεμήσουμε την τρομοκρατία και τον βίο εξτρεμισμό. Ελπίζω ότι αυτή η ενότητα θα μεταφραστεί σε συνένεση στο Συμβούλιο και μεταξύ των θεσμικών οργάνων θα πρέπει να αυξήσουμε τις προσπάθειες να κρυζώσουμε την τρομοκρατία της κοινωνίας μας. Οι βελικές αρχές απέτρεψαν τρομοκρατική συνωμοσία την περασμένη εβδομάδα και βλέπουμε ότι η τρομοκρατία ότι μπορεί να ξεμητήσει οπουδήποτε, ποτεδήποτε. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η εσωτερική ασφάλεια και οι μυστικές υπηρεσίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Στην Προεδρία μα θα υποστηρίξουμε τι προσπάθειε των κρατών μελών να αυξήσουν την καταπολέμηση τη τρομοκρατία, σχετικέ επιχειρήσει και να συντονίσουν τι επιχειρήσει. Άρα πρέπει να χρησιμοποιούμε τα υπάρχοντα μέσα και να εφαρμόσουμε πλήρω τη στρατηγική καταπολέμηση τη τρομοκρατία και την καταπολέμηση των ξένων μαχητών. Στην του Παρισίου των Παρισίων στις 11 ε, Ιανουαρίου συμφωνήσαμε να διευρύνουμε τη συνεργασία και να αυξήσουμε την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Άρα θα πρέπει να προωθήσουμε τα στοιχεία των επιβατών που θα πρέπει να συλλέγονται και να επιβάζονται, θα πρέπει να δικοποιήσουμε ε, την, την προστασία μας εναντί των, και τα μέτρα όσον αφορά τις χώρες προέλευσης. Να καταπολεμήσουμε την διαμόρφωση ριζοσπαστικών θέσεων, τη χρηματοδότηση αυτών, και θα πρέπει το διαδίκτυο να μην χρησιμοποιείται για τη στατολόγηση τρομοκρατών. Θα πρέπει να συνεργαστούμε πιο στενά με τους διεθνείς συμμάχους μας όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Αυστραλία και, να και θα πρέπει να προωθούμε στο διάλογο Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτε χώρε τα θέματα καταπολεμή τρομοκρατία και θα παρουσιάσουμε νέα στρατηγική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την εξωτερική πολιτική. Προσβλέπουμε στι προτάσει που είναι ένα τμήμα του πακέτου καταπολεμήσεω των τρομοκρατών, τη τρομοκρατία ερήτημα μέλη. Πάμε στη διεύρυνση τώρα. Θα εστιαστούμε τώρα σε σημαντική ε, πτυχή που είναι η συμμετοχική ε, Ευρώπη, που είναι στο πρόγραμμα της Προεδρίας. Στο επόμενο εξάμεινο ελπίζουμε να προωθήσουμε τις διαπραγματεύσεις όπου αυτό είναι εφικτό. Δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν μεγάλες πολιτικές ευαισθησίες σε πολλά κράτη-μέλη καθώς και ότι ε, οι μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται είναι πολύ δύσκολες. Θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι η διεύρυνση ήταν το πιο αποτελεσματικό εργαλείο εξωτερική πολιτική. Η διεύρυνση αύξασε την ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή, οδηγεί σε ευημερία σε όλη την Ήπειρο. Και δίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θέση πολύ μεγάλη στο διεθνέ προσκήνιο. Η προπτική ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει κίνητρα για πολιτικέ μεταρρυθμίσει, οικονομικέ μεταρρυθμίσει, αλλάζει τι κοινωνίε. Σίγουρα αυτό ίσχυσε στην Λετωνία και στι άλλε βαλτικέ χώρε τη δεκαετία του 90. Η διεύρυνση διαδίδει τις αξίες Ευρώπης και τα πρότυπα και εκτός συνόρων και όχι μόνο σε εκείνους που γίνονται μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσης τελικά. Μπαίνουν κάποιες χώρες και άλλες θέλουν να μπουν. Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις εξακολουθούν να εδράζονται επί της αξίας των χωρών και επί αιρεσιμότητας, επί μαθημάτων που μάθαμε από τις πρώτερες διευρύνσεις. Οι χώρες κρίνονται κατά περίπτωση και και προδεύουν οι συνομιλίε ταχύτερα άμα οι μεταρρυθμίσει προχωρούν πιο γρήγορα. Αν πληρούνται τα κριτήρια τη Κοπενχάγη και το κράτο δικαίου και τα πρότυπα για την οικονομική διακυβέρνηση και για την δίκηση, ε, τότε επιταχύνουν τη διαδικασία. Η μεταρρύθμιση δεν είναι κάτι απλό. Έχουμε θέσει ψηλά τον πύχη, αλλά αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Θέλουμε να διαδώσουμε τι αξίε μα και όχι να τι αποδυναμώσουμε, να μοιραστούμε τι επιτυχίε μα και να μην περιορίζουμε τι επιτυχίε και να ενισχύσουμε την Ένωση. Θα πρέπει όμως επίσης να είμαστε και συνεπείς, άρα θα πρέπει να ανταμείβουμε την πρόοδο όταν αυτό πρέπει κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Ελπίζουμε να είμαστε σε θέση να προωθήσουμε τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Θέλουμε να πετύχουμε πρόοδο στις συνομιλίες με τη Σερβία και ελπίζουμε τελικά να ανοίξουμε τα πρώτα κεφάλαια κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Αυτό θα εξαρτάται από την πολιτική βούληση του Βελιγραδίου, από πρόοδο όσον αφορά το κράτο δικαίου και την εφαρμογή των επιτευθέντων συμφωνιών ε, στι συνομιλίε του επίπεδου με την Πιστίνα. Σταδιακή εξομάλυνση των σχέσεων θα πρέπει να επιτρέψει και περαιτέρω πρόοδο όσον αφορά τη σταθεροποίηση και τη συμφωνία σταθερότητα και σύνδεση με το Κωσυφοπίδιο που ελπίζουμε να υπογραφεί το πρώτο εξάμεινο του 2015. Παρομοίω προσβλέπουμε στη συνέχιση ενταξιακών διαπραγματεύσεων με το Μαυροβούνιο και να ανοίξουν και νέα κεφάλαια. Καλωσορίζουμε τη δέσμευση του Μαυροβονίου για να κινηθεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πρόοδο την επιτευχθήσα όσον αφορά τη διάφορε που χρειάζονται περισσότερα για το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Θέλουμε να υποστηρίξουμε την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με την Άγκυρα. Η Τουρκία είναι στρατηγικό μα εταίρος, με την οποία έχουμε κοινά συμφέροντα και κοινέ προκλήσεις. Ελπίζουμε το παρόν πολιτικό πλαίσιο δεν είναι ευνοϊκό, όμως πιστεύουμε ότι οι δεξιακές διαπραγματεύσεις είναι το καλύτερο πλαίσιο για τη σχέση Ευρωπαϊκής Ενώσεως Τουρκίας και είναι ο μηχανισμός για την ενθάρρυνση μεταρρυθμίσεων. Παρ' όλα αυτά παροτείνουμε την Τουρκία να αποδείξει σαφώς ότι θέλει να ενστερνιστεί τις ευρωπαϊκές αξίες. Δεν υπήρξε ομοφωνία όσον αφορά τι δεξιακέ διαπραγματεύσεις με το ΦΥΡΟΜ τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του περασμένου Δεκεμβρίου αναφέρονται στη δυνατότητα να επαναξεταστεί το θέμα το 2015. Ένα θετικό μήνυμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα παράσχει ενθάρρυνση και για τη ΦΥΡΟΜ και την ευρύτερη περιοχή. Όμως το ΦΥΡΟΜ θα πρέπει να δείξει ότι έχει πολιτική βούληση και να συνεχίσει την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Ε, έχουμε ε, η Σλοβενία ε, αναγνωρίστηκε ότι είχε γίνει πάρα πολύ σκληρή δουλειά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλωσορίζουμε την πρόοδο που έχει επιτεθεί, αλλά περισσότερες προκλήσεις ε, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν πριν να ανοίξουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Εν τω μεταξύ ανησυχούμε για την αποτελμάτωση όσον αφορά την Βοσνία Ζεγοβίνη. Θέλουμε να γίνουν ε, μεταρρυθμίσεις Είμαι πραγματιστής για τα εμπόδια, πιστεύω όμως ότι στην Προεδρία μας μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο διαπραγματεύσει με τις υποψήφιε χώρες και όσον αφορά το Σύμφωνο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με τα Δυτικά Βαλκάνια. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε άλλα θέματα που τίθενται για την Επιτροπή σας ε, όσον αφορά τις σχέσεις με την Ελβετία. Η Ελβετία είναι σημαντική εταιρεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικό να συνεχιστούν οι συνομιλίε όσον αφορά το διοργανικό πλαίσιο για τι σχέσει μεταξύ Ελβετία και Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Σεβόμαστε τα αποτελέσματα του στην Ελβετία, όμω θέλουμε ελεύθερη διακίνηση προσώπων ή θεμελιώδου σημασία για την ευρωπαϊκή πολιτική. Η εσωτερική αγορά, οι τέσσερι ελευθερίε ε, υποστηρίζονται. Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με την Ελβετία θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της ε, συμφωνίας Αξιότιμα μέλη, η διεύρυνση είναι μία από τις προτεραιότητες για την ε, συμμετοχική Ευρώπη. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και την Προεδρία μας για να προχωρήσει σε άλλους τομείς η Ευρώπη. Να προωθήσουμε την ειρήνη και σταθερότητα στην γειτονία μας, στην Ουκρανία, τη Λιβύη και τη Συρία. Θέλουμε να στηρίξουμε το έργο όσον αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία. Ε, στη Ρίγα θα γίνει το Μάιο για την Ανατολική γειτονία και θέλουμε να προωθήσουμε και θέματα μετανάστευση. Κεντρική Ασία θέλουμε να γίνουν προσπάθειες αναθεώρησης των σχέσεων και θέλουμε να προωθήσουμε τις σχέσεις, ε, τη στρατηγική Ευρωπαϊκής Ενώσεως για την Κεντρική Ασία, να ενθαρρύνουμε το εμπόριο, συμφωνίες με τον Καναδά, την Ιαπωνία και με τη ΣΥΠΑ όλος ιδιαίτερος. Και είναι πάρα πολύ ευχάριστο για μένα το να μπορούσα να μιλήσω σήμερα εδώ και ενδιαφέρον πάρα πολύ να ακούσω τις απόψεις και να απαντήσω τις ερωτήσεις. Κύριος Πρέντα, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε που ήρθατε να μας δείτε και να μας παρουσιάσετε τις προτεραιότητες της Λετωνικής Προεδρίας. Στο ίδιο πνεύμα έκανε ο Πρωθυπουργός της χώρας σας την ε, σχετική παρουσίαση στην Ολομέλεια πριν από μια εβδομάδα και συγχαρητήρια για τις ε, φιλόδοξες προοπτικές σας. Σας εύχομαι καλό κουράγιο και όλα αυτά τα οποία είπατε πειράζονται πάρα πολύ από τις τρομοκρατικές απόπειρες που σημειώθηκαν. Κάτι σε σχέση με την Ερζεγοβίνη, γιατί έχω αναλάβει μια σχετική έκθεση για την χώρα αυτή. Επίσης, σήμερα μόλις συζητήσαμε δύο εκθέσει για Κοσμοπέδιο και Σερβία. Τον επόμενο μήνα θα συζητήσουμε και για την Βοσνία. Και εσείς τι θεωρείτε, ότι θα υπάρξει κάποια σημαντική πρόοδος κατά την Προεδρία σας ή θεωρείτε ότι το επόμενο εξάμεινο θα έχουμε απλώς έναν συντονισμό και από τη μία μεριά θα έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη μεριά θα έχουμε τις προσπάθειες ε, Αμερικανών, ε, ίσως και Βρετανών ε, για να εξευρεθεί τελικά ένας τρόπος, κάποια μέσα ούτως ώστε να μπορέσουμε να διεκπαιρεώσουμε τα θέματα αυτά πριν το τέλος της Προεδρίας σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπουργέ, σας χαιρετίζουμε εδώ στο Κοινοβούλιο και ελπίζω ότι η Προεδρία σας θα στεφτεί με επιτυχία. Έχω μία ερώτηση. Την προηγούμενη Παρασκευή στη Λετωνία εκλήθησαν ε, οι κάτοικοι να μιλούν λετωνικά μόνο. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα εσωτερικό σχόλιο. Ήταν εσωτερικό αν θέλετε. Δεν ήταν θέμα εξωτερικής πολιτικής. Αλλά ποια είναι η δική σας άποψη. Πώς πιστεύετε ότι τέτοιες ε, πολιτικές σε συνάδουν με την ε, επίσημη εξωτερική πολιτική της Λετωνίας όπου ξέρουμε ότι στη Λιτωνία και σε όλη την Ευρώπη υπάρχει, υπάρχουν ε, ε, διεθνείς σχέσεις και αυτό έχει και για την Αρμενία, τη Λευκορωσία. Πώς λοιπόν εκτιμάτε εσείς την κατάσταση. Είσαστε πρόεδρος από την χώρα που κατέχει την Προεδρία. Πώς ε, είναι η στάση σας λοιπόν σε ό,τι αφορά τις εθνικές μειονότητες στην Ευχαριστώ. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε, Υπουργέ, στην Επιτροπή. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία επευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων σας. Κάθε επιτυχία σας εύχομαι ασφαλώς. Επιτρέψτε μου να σας ε, κάνω μια σύντομη ερώτηση. Υπάρχουν ε, εξαιρετικά ενδιαφέροντα όργανα, υπηρεσίες στην Λετωνία, στην Ρήγα. Ακούσαμε την έκθεση στην ε, συνέλευση του ΝΑΤΟ σε ό,τι αφορά τη Ρωσία. Θα ήθελα να εστιαστώ σε θέματα προπαγάνδας από πλευράς της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της Δύσης. Πώς ε, σκοπεύετε να αξιοποιήσετε την εμπρογνωμοσύνη τέτοιων κέντρων προκειμένου να εξουδετερώσετε αυτές τις απόπειρες κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων δυτικών εταίρων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ερώτηση προς την Υπουργή Εξωτερικών. Κάτι για τη Συμφωνία του Μίνσκ που δεν εφαρμόστηκε και επομένω δεν υπάρχει ουσιαστικά στην Ανατολική Ουκρανία εκεχηρία και κατάπαυση πυρό. Εσεί κατά την προεδρία σα, τι μπορείτε να κάνετε ούτω ώστε η συνθήκη του Μίνσκ να εφαρμοστεί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, και εγώ να σας ευχηθώ ότι καλύτερο, καλώς ορίσατε. Και όσον αφορά τις πληροφορίες για τους συμβάσεις των αεροπορικών εταιριών, το PNR, είναι πολύ σημαντικό. Θα σας δείξω κάτι, να μου πείτε για την εταιρική σχέση προς Ανατολάς. Έχουμε έξι χώρε που εκεί συμμετέχουν. Από αυτέ τι έξι, τρει έχουν συμφωνία σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι βρίσκονται σε πιο προχωρημένη φάση από τι υπόλοιπε. Άλλε δύο χώρε και από αυτέ έχουν ε, συνάψει την Ελληνική Ένωση. υπάρχει και μια χώρα, το Αζερβαϊτζάν, το οποίο ας πούμε ότι είναι ουδέτερο, δεν μπορώ άλλο χαρακτηρισμό. Τώρα, πέραν της συμφωνίας της Ρήγας, πέραν των πρακτικών αναθεμάτων, απορρίθμιση κλπ. Θεσμικά, τι άλλη πλαισίωση φαντάζεστε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε σε αυτήν την συνεργασία προς Ανατολάς, την εταιρική σχέση προς Ανατολάς, Thank you very much, Ο κύριο ευχαριστώ πολύ. καλώ ορίσατε κύριε Υπουργέ. Σα είδαμε και με του συντονιστέ. Πάρα πολύ θετικό αυτό το οποίο κάνετε, συνεργαστούμε. Ελπίζουμε και όπω είδατε και στην αρχή, έχετε κατά τη τρομοκρατία, έχετε και άλλε προκλήσει να αντιμετωπίσετε και βεβαίω θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα προδικάζουμε το τι, πώς θα εξελιχθούν τα πρώτα, θα κάνετε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και λοιπά, όλες αυτές τις ευθύνες ε, που έχετε αναλάβει για εσωτερικό και εξωτερικό. Οπότε καλή πτυχία για όλες αυτές τις προκλήσεις. Και συμφωνώ σε όσα είπατε για την Ρωσία. Η πολιτική μας ομάδα θέλει να βελτιωθούν οι σχέσεις με την Ρωσία. Βλέπουμε ότι εκεί υπάρχουν ευκαιρίες θετικό διάλογο. Όμως δεν πρέπει να αγνοήσουμε την σωρία παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου. Θα πρέπει κάτι να κάνουμε για την κρίση στην Ουκρανία, αλλά πρέπει να δούμε και για τον ρόλο της Ρωσίας στην Συρία που και αυτό είναι σημαντικό για μας. Έχω δύο ερωτήσεις πολύ σημαντικό ο ρόλο σας στο εσωτερικό της χώρας σα πέραν της προεδρίας που ασκείτε. Πέστε μας, αν θέλετε, για την Λετωνία, τι γίνεται με τους ε, ΛΟΑΔ. Για την πολιτική μα ομάδα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και για όλους τους Ευρωπαίους, γιατί υπάρχει προβληματισμός. Γιατί κάποιοι από την κυβέρνησή σα έχουν κάνει κάποιε ανησυχητικέ δηλώσει όσον αφορά το τι γίνεται για το κατά πόσον θα επιτρέψετε να ασχοληθούν κάποιοι ΛΟΑΔ σε θέσεις ε, ε, της υπηρεσίας εξωτερικής Επίσης, και σήμερα είπαμε ότι έχουν γίνει κάποιες συνεντεύξεις και επειδή αυτό πρέπει να γίνεται στην γλώσσα σας. Θα πρέπει πάντως να σεβαστείτε τον πλουραλισμό, να σεβαστείτε τις μειονότητες. Να, ποιο μήνυμα μπορείτε να στείλετε στην Ρωσία. Hvala lijepa. Eh, gospod ministar, Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Πριν από κάποια χρόνια ήμουνα ο πρώτος ε, Σλοβαίνος πρέσβης στη Λετωνία. Κύριε Υπουργέ, σήμερα μιλήσαμε για την πρόοδο που έχει σημειωθεί από πλευρά των υποψηφίων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι μόνιμος συζητητής για την πρώην Κυκλοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η χώρα μου έχει αναγνωρίσει την χώρα αυτή υπό το όνομα Μακεδονία, γι' αυτό έτσι θα ήθελα να συνεχίσω να την αναφέρω. Αναφέρατε σκεπτικότητα και σε ό,τι αφορά σκεπτικισμό, σε ό,τι αφορά τη σχέση σας με τη σχέση μας με την Νέα Μακεδονία. Δεν συμφωνώ με την άποψή σα Από όλε τι υποψήφιε χώρε. η Μακεδονία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο θεωρώ ότι εφαρμόζει το κοινωτικό κεκτημένο. Το πρόβλημα προκύπτει από το ατυχές αυτό περιστατικό από την, από τη διαφωνία με την γειτονική χώρα σε ό,τι αφορά το θέμα της ονομασίας. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ το συντομότερο δυνατόν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις ενώ το Συμβούλιο θα πρέπει να σταματήσει να παρεμποδίζει τις διαπραγματεύσεις. Η ανάληψη των διαπραγματεύσεων μπορεί να οδηγήσει σε επίλυση των εκτών ζητημάτων, όπως μεταξύ άλλων και το θέμα του ονόματος. Σας απευθύνω έκκληση λοιπόν εδώ να διατραματίσετε ενεργό ρόλο στο θέμα αυτό. Το κράτος αυτό μπορεί να επηρεάσει τη σταθερότητα της όλης ε, περιοχής. Μία δεύτερη ερώτηση. ως ε, ηγέτη σε θέματα πολιτικής εξωτερικής, ε, εξωτερικών υποθέσεων τα επόμενα έξι μήνες, επόμενους έξι μήνες. Μπορείτε να αγγιηθείτε ότι στα κράτη όπου δεν γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα θα διατεθούν όλα τα μέσα που υπάρχουν Έχω κατά νου το Μαρόκο, το Ισραήλ, την Τουρκία και πολλά άλλα κράτη. Σα ευχαριστώ, συνάδελφοι. Θα ήθελα να σα παρακαλέσω, επειδή έχουμε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι η συζήτηση για την διαβρυνσή να επικεντρωθείτε σε θέματα Ουκρανία, Ρωσία, στα θέματα των και στι ερωτήσει που έχουν να κάνουν με το συγκεκριμένο τμήμα. Σα παρακαλώ λοιπόν να επικεντρωθείτε στα θέματα διεύρυνση, λέει ο Προεδρο. Το λόγο έχει τώρα ο συνάδελφο Μιλαμών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ που ήρθατε. τι καλύτερε ευχέ μα για την Προεδρία. Που αυτόν τον μήνα ξεκινά. Στο τέλο τη ήγησης σα είπατε πόσο σημαντικέ είναι οι συμφωνίε με τι ΗΠΑ και Καναδά με τον Καναδά ουσιαστικά έχει τελειώσει η πόρη αυτή. Θα πρέπει τώρα η Επιτροπή μάλιστα να δώσει μια τελευταία όθηση και έτσι να έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδρομή στο τέλος του έτους. Αλλά πρέπει, πρέπει και εσείς να δώσετε μια όθηση. Τώρα, όσον αφορά τη ΣΥΠΑ και την Αμερικανική πέρα, έχουμε τον Ιούνιο συνάντηση κορυφής με την ΣΕΛΑΚ Οπότε θα πρέπει με την ευκαιρία αυτή, με τη Λατινική Αμερική, να συσφίξουμε τις σχέσεις, γιατί έχει σημασία αυτή η περιοχή. Άρα, είναι σημαντικό αυτό το εξάμεινο για τις σχέσεις Ευρώπης με όλη την Αμερικανική Ήπειρο. Ačiū gerbiamas και e, gerbiamas ministrė. Aš taip Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Επικέ. Θα ήθελα και εγώ να σας συγχαρώ, να συγχαρώ Τριτονία για την ανάληψη των καθηκόντων της. Ε, όλοι ελπίζουμε στα βέλτιστα αποτελέσματα. Αναφερθήκατε στα θέματα διεύρυνσης. Αναφερθήκατε στην ε, περίπτωση της Τουρκίας. Έχετε ελπίδος ότι θα ξεκινήσει να κινείται η κατάσταση σε σχέση με την σημερινή κατάσταση. Αναρωτιέμαι κατά πόσον η Λετωνία θα είναι το κράτος που θα σημειώσει τη σημαντική πρόοδο στο θέμα της ε, διεύρυνσης και στο θέμα της τουρκικής προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Thank you, Chairman. Mr. Minister. Ευχαριστώ, Πρόεδρε Υπουργέ. Σας ευχόμαστε ότι καλύτερο για την ε, Προεδρία σας και σίγουρα θα είναι πολύ άσχολη και πολύ σημαντική η επόμενη περίοδος για όλους. Ελπίζουμε να μπορέσετε τα καθήκοντα να τα εκπληρώσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Υπουργέ, στον τύπο είδαμε την πρόθεσή σας να μεταβείτε στη Μόσχα για διαπραγματεύσεις με τον κ. και με την ηγεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Υπουργέ, τι είδου μήνυμα θα διαβιβάζετε στη Μόσχα Και σίγουρα φαντάζομαι θα αναφέρετε την ρωσική επίθεση στην Ουκρανία. Σήμερα λάβαμε την πληροφορία ότι δύο στρατεύματα 700 μέχρι 700 άτομα ε, πέρασαν τα σύνορα με την Ουκρανία. Θα εκτιμούσα λοιπόν σχολιασμό της κατάστασης στην Ουκρανία από πλευρά σας. Thank you. Herr Chairman. On the enlargement in the Western Balkans, Mr. Minister, thank you very much for your... Ευχαριστώ για τη διεύθυνση Δυτικά Βαλκάνια. Καλά τα εισαγωγικά σας σχόλια. Εξέλαβα ότι θέλετε να χρησιμοποιήσετε την εμπειρία σας από τις ταξιακές διαπραγματεύσεις και στηρίζω την απλή γλώσσα που χρησιμοποιείτε που μαρτυρά ότι θέλετε να πετύχετε κάτι θέλετε να προωθήσετε τα πράγματα από την παρούσα κατάσταση τα, τα επόμενα πέντε χρόνια δεν θα υπάρξει διεύρυνση, διότι αντικειμενικά καμία από τις υποψήφιες χώρες δεν θα είναι έτοιμη για, έτοιμη, συγγνώμη, για την ένταξη. Ε, ξέρετε όμως ότι είναι απαραίτητο η ορολογία να χρησιμοποιείται σωστά, με πολύ ευαισθησία. Διότι οι δηλώσεις του Προέδρου Γιούνκερ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ανησύχησε πολύ τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, τους εταίρους μας. Εκτιμώ λοιπόν την προσέγγισή σας. Γνωρίζω ότι γνωρίζετε τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Δύσκολο να εφαρμόσετε αυτά που θέλετε. Είναι φιλόδοξη η στόχοι που θέσατε και αναφέρατε. Αλλά αξίζεται την υποστήριξή μας και τη βοήθειά μας για να είστε επιτυχείς θα πρέπει να συνεργαστείτε στενά με την ύπατη εκπρόσωπο Μογκερίνη, με την υπηρεσία εξωτερική δράση, με του επικεφαλεί των αντιπροσωπείων στις χώρες αυτές. Ερώτηση. Ποιες είναι, ποιες είναι οι καλύτερες προσεγγίσεις όσον αφορά τις επαφές για να πετύχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ συζητώντας τρόπους για να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία. Συζητήσατε την ανάγκη για περισσότερα χρήματα για να επενδυθούν αυτά όσον αφορά την ε, ασφάλεια των μυστικών μας υπηρεσιών και καλύτερο τρόπο διαβίβασης πληροφοριών των μεταξύ μυστικών υπηρεσιών, κάτι που δεν υπάρχει. Να επενδύσουμε σε προγράμματα για την αποφάση Φυγή της, ε, του προσελητισμού των νέων προς ε, ακραίες θεωρίες. Στην πρώτη γραμμή καταπολεμής τρομοκρατία στο Ιράκ. Επέστρεψα τώρα με συναδέλφους και είδα ότι δεν υπάρχει Ευρώπη εκεί. Τα κράτη-μέλη δεν συντονίζουν και την παροχή όπλων καν προς τους Πεσμέργα δεν υπάρχει συντονισμός μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια με την ΕΚΟ. Δεν υπάρχει συντονισμός ανθρωπιστικής βοήθειας σε σχέση με την αναπτυξιακή βοήθεια. Και δεν έχουν σχολεία οι πρόσφυγες που να λειτουργούν. Μιλώ για τα στρατόπεδα, για τους Γιαζίδη και τους χριστιανού. χριστιανούς. Ε, δεν υπάρχουν προγράμματα για την απελευθέρωση των απαχθέντων στρομοκράτες. Δεν υπάρχει πρόγραμμα να βοηθήσουμε τις ε, γυναίκες Αζίδη που ε, έχουν γίνει σκλάβοι, σκλάβες των τρομοκρατών. Ε, και αυτό θα πρέπει να το συντονίσουμε με τους ντόπιου. Το ίδιο θα μπορούσα να πω και για τη Λιβύη, που έχει γίνει καταφύγιο τρομοκρατών. Πού είναι η Ευρώπη? Myself. Λιβύη, Ουκρανία, τρομοκρατία είναι στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων και θα αναφερθούν σε επόμενη έκθεση. Εδώ μιλάμε για τη διεύρυνση. Πλένκοβιτς, επόμενος συνάδελφος που έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Εγώ συμμετέχω στην αντιπροσωπή για την Ουκρανία. Ό,τι με ενδιαφέρει να πείτε τι θα κάνετε το ξένο της Προεδρίας, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε πιο συνεπείς, συνεκτικές ε, διπλωματικές ενέργειες ως Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο ώστε να καταλήξουμε για το Ντόμπας ε, ε, με μια λύση, αλλά να δούμε και με την παράνομη προσάρτηση της ε, Κρυμαίας. Τώρα, όσον αφορά την διεύρυνση, νομίζω ότι είναι σημαντικό το ότι τονίσατε τα βασικά σημεία για την πιο πρόσφατη προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε και εμείς θα πρέπει ε, να παρακολουθήσουμε τη συνέχεια αυτής της πορείας κατά την παρούσα θητεία του Κοινοβουλίου. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, και εγώ να σας καλωσορίζω τι καλύτερες ευχές για την Προεδρία της χώρας σας. Μας μιλήσατε για την διεύρυνση, μιλήσατε για την Τουρκία είπατε ότι πρόκειται για στρατηγικό εταίρο. Εγώ θέλω τώρα να αναφέρω την Βοσνία και την πρώτη που έχει σημειωθεί. Αν θέλετε, πες μας δυο λόγια. Τώρα, όποτε θέλετε, τι γίνεται με την τρομοκρατία. Πώς είναι να τον καλύψουμε, να πλησιώσουμε τους μουσουλμάνων. Υπάρχει μεγάλη ελεξάρτηση στο σημερινό κόσμο. Επίσης, όλο ένα και περισσότερες επιθέσεις σημειώνονται κατά των μουσουλμάνων. Τι μπορεί να κάνει η Προεδρία σας. Mr. Chairman. Minister, first I would like to... πρώτα πρώτα καλή επιτυχία, Πρόεδρε. Προς τον κύριο Υπουργό και αυτό που θέλω να ρωτήσω αφορά 100% την ε, διεύρυνση. Ξέρετε ότι από την Αλβανία έχουμε καλά μαντάτα. Θεωρείτε ότι εάν συγχυστούν ε, αυτά τα θετικά βήματα μπορεί να ανοίξει κάποια κεφάλαια διαπραγματευτικά η Αλβανία κατά την ε, Λετωνική Προεδρία. Κάτι άλλο τώρα. Η Ισλανδία. Έχουμε τώρα δύο τάσεις στη χώρα. Πρώτα-πρώτα ο κυβερνητικό εσπισμό θέλει να κάνει ένα δημοψήφισμα για να σταματήσουν οι διαπραγματεύσει. Όμω οι σοσιαλδημοκράτε θέλουν να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσει. Εάν έχουμε και μια κυβέρνηση, αν δεν γίνει τέτοιο δημοψήφισμα, προτίθεστε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσει με την Ισλανδία. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρο θέλω να ξεκινήσουμε τώρα το κομμάτι κυκλισμένο των θυρών και θα μπορέσουμε να συνδέσουμε αν τα δύο κομμάτια όσο πιο επικοδομητικά